Καλησπέρα σας. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής TEX 3. Έχοντας ακούσει εμπειρογνώμονες, επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και υπουργούς κατά το πρώτο οκτάμινο της εντολής της TEX Τρία, οι συγκητές θα παρουσιάσουν σήμερα τα απορίσματά τους και τις συστάσεις περί βελτιώσεως του ενωσιακού πλαισίου στην καταπολέμηση του φαινομένου του ξεπλήματος χρήματος και της διαφθοράς. Η αγγλική εκδοχή του σχεδίου εκθέσεως δυναμήθη στα μέλη στις 14 ε, Νοεμβρίου. Όλες οι γλωσσικές εκδοχές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Text 3 της Επιτροπής. Το χρονοδιάγραμμα ως εξής. Προθεσμία για αποβολή τροπολογιών στις 5 το απόγευμα της 17ης Δεκεμβρίου συζήτηση των τροπολογιών 29 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 27 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους και ψηφοφορία και συζήτηση στην Ολομέλεια στη δεύτερη σύνοδο του Μαρτίου στο Στρασβούργο του χρόνου. Και οι δύο συνεισηγητές θα έχουν 7 λεπτά ο καθένας για εισαγωγές και μετά τετράλεπτες παρεμβάσεις των σκιωδών εισηγητών θα ακολουθήσουν και μετά θα λάβουν το, χώ, το λόγο άλλοι ομιλητές. Ο εισηγητής του ΕΛΚ, ο κ. Νταμάη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς χαίρομαι που έχω λιγότερα λεπτά στη διάθεσή μου από τα μέλη. Έχω περισσότερα από ότι τα μέλη. Δεν θα χρησιμοποιήσω και τα 7 λεπτά. Πριν από πολλά χρόνια ξεκινήσαμε την, αυτή την ειδική επιτροπή και η κατάσταση εξελίχθηκε στις εργασίες τεσσάρων ειδικών επιτροπών και μια επιτροπής τη ΕΚΟΝ. Και φαίνεται ότι η καταπολέμηση των παρανόμων εσόδων, της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγή και η προσπάθεια μεγαλύτερη δικαιοσύνη στη φορολογία και τη διαφάνεια είναι κάτι που δεν έχει λήξει. Αυτό αποδεικνύεται και από πρόσφατα σκάνδαλα όπως τη ΚΑΜΕΞ. Η έκθεσή μας συνοψίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το πρώτο σκάνδαλο και την πρώτη συνεδρίαση των Lux Leaks το 2015 μέσω των εργασιών άλλων των επιτροπών της τάξε, της τάξε 2 και της ΠΑΝΑ και εξετάζουμε ποια κενά απομένουν, ποιες αδυναμίες του συστήματος παραμένουν και που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από προβλήματα στα διάφορα πεζικά σκάνδαλα και στην Κάμεξ, στο σκάνδαλο Κάμεξ, προοδεύουμε, θα έλεγα, σε πολλούς τομείς και θα πρέπει να είμαι θα υπερήφανοι για τα επιτεύγματα και έχει παίξει σημαντικό ρόλο το Κοινοβούλιο σε αυτά. Έχουμε νέα νομοθεσία, έχουμε αυξήσει τη διαφάνεια σε πολλούς ε, τομείς και υπάρχει αυξανόμενη προθυμία για αντιμετώπιση των προβλημάτων σε πολλούς τομείς. Εξακολουθούμε να μην έχουμε θάρρος και κοινή προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με καλύτερο τρόπο μαζί όπως το CCTP και τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ. Και είναι αρκετά σαφές ότι σε άλλε πτυχέ δεν λείπει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο όπως το ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας, υπάρχει έλλειψη συνεργασίας και αυτά υπονομεύουν το αποτέλεσμα. Επίσης, εγώ θα έλεγα ότι εν γέννη και συνολικά και το είπα λυπούμενος ότι υπάρχει απροθυμία από τα κράτη-μέλη να απεμπολίσουν ένα μικρό τμήμα κυριαρχίας ούτως ώστε να μπορέσουν να πολεμήσουν αποτελεσματικά τα παρόντα προβλήματα. Δεν έχουν αυτή τη βούληση και αν δεν αλλάξει αυτό δεν θα προχωρήσουμε πιθανότατα στην έκθεση. Έχουμε καλύψει πάρα πολλά θέματα, ευρύ φάσμα θεμάτων. Να τονίσω ότι ήμασταν περιορισμένοι από το πεδίο εφαρμογή και γι' αυτό έχουμε ετοιμάσει διάφορες τροπολογίες που θα υποβληθούν αργότερα. Ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε, βλέπετε, όλα τα σημαντικά στοιχεία θα καλύπτονται. Θα ήθελα να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη να μην κουβεντιάζετε μεταξύ σας. Να αρχίσω από την αρχή, λέει ο Α, ίσως και όχι. Λοιπόν, αυτό που βλέπω σαν εστιακό σημείο της εκθέσεως που ίσως δεν είχα προσεχθεί κατά το παρελθόν είναι το ξέπλυμα χρήματος, οι απάτες του ΦΠΑ και κάποια συγκεκριμένα προβλήματα όπως η χρυσή θεώρηση, η χρυσή βίζα τονίζουμε και κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι φορολογικές και άλλες αρχές έχουν ισχυρά εργαλεία διαθέσιμα και πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία και έπρεπε να εστιαστούν σε αποτελεσματική χρήση και ε, διαβίβαση αυτών πληροφοριών. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερε εξουσίε και δυνάμει και περισσότερα στοιχεία, αλλά χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερη χρήση των υπαρχόντων στοιχείων. Ε, κατά παρελθόν εστιαζόμεθα στην εξάλληψη της διπλής φορολόγησης, αλλά θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα της διπλής φορολογήσεως των φορολογουμένων, της αυξήσεως του κόστους, το άχθος, ε, συμμορφώσεως με τις φορολογικές υποχρεώσεις και η αβεβαιότητα που περιβάλλει την υποχρέωση καταβολής των φόρων, θα πρέπει και αυτά να τονιστούν, διότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε δίκαιη και αξιοπιστή οι δίκαιοι και αξιοπρεπεί και ειλικρινεί φορολογούμενοι να βραβεύονται την ειλικρινιά του. και εμείς να επικεντρωνόμαστε στον κυνηγάμε του κακούς. Στον τομέα της καταπολεμήσης του ξεπλήματο χρήματο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα είναι πραγματικά στεναρό, ισχυρό. Αν τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν σωστά την νομοθεσία, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο η οδηγία κατά πολέμηση του ξεπλήματο χρήματο μήπω θα πρέπει να μεταμορφωθεί σε κανονισμό για να βελτιώσουμε τη σαφήνεια και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει καλύτερη επιβολή τη νομοθεσία. Θα μπορούσα να μιλήσω περισσότερο, αλλά και ο ΓΕΠ θα ήθελε να αναφερθεί στα δικά του σημεία. Θέλω να τον ευχαριστήσω για επικοδομητική συνεργασία που είχαμε, που ελπίζω θα συνεχιστεί. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε το ότι το μήνυμα που θα προέλθει από αυτό το κοινοβούλιο στον τομέα αυτό θα είναι σαφές και ότι δεν σταματήσει το έργο μας και θα συνεχιστεί. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση του έργου σας κύριε Πρόεδρε, ε, της Γραμματείας και των άλλων μελών της Επιτροπής. Ήταν πραγματικά κάτι που μας βοήθησε πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γεπε του του τους για 7 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω τον Λούντι Λούντικ Νίντερμαϊρ για την επικοδομητική του συνεργασία. Απόλαυσα την έκθεση αυτή. Δεν είναι μυστικό ότι διαφωνούμε σε αρκετά πράγματα, αλλά καταφέραμε να βρούμε κάποιους συμβασμούς στα περισσότερα πράγματα και μια συμφωνία κύριων. Συμφωνήσαμε να διαφωνήσουμε σε άλλα. Επίσης ε, δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω την ε, γραμματεία και την ομάδα του Λούντεκ ε, και των σοσιαλδημοκρατών. Πραγματικά απαιτήθηκε φοβερή προσπάθεια από όλους μας. Τώρα εγώ θεωρώ ότι η δουλειά αυτή έχει αποτελέσματα. Νομίζω το ανέφερε και ο Λούντεκ. Τώρα έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης ε, το οποίο είναι αρκετά λεπτομερές, ε, σαφές ε, και ξεκάθαρο. Δεν διστάσαμε να κατονομάσουμε χώρες, εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν ανταποκριθήκαν στις ευθύνες τους και ακριβώς είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά στην Επιτροπή και στο κοινό. Ταυτόχρονα αυτό το κάνουμε μόνο εκεί όπου είναι τεκμηριωμένο. Και ακριβώς έχει μεγάλη σημασία αυτό. Μπαίνουμε σε λεπτομέρειες των μεγαλύτερων υποθέσεων ξεπλήματος χρήματος που αποκαλύφθηκαν στην θητεία της Επιτροπής μας και πάλι βασισμένη σε γεγονότα. Προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις για τους ελεύθερους λιμένες, τις ειδικές οικονομικές ζώνες, τα patent box, ενίσχυση των θεσμικών οργάνων, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και παγκόσμια δράση υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε και αναψώμενες χώρες να είναι μέρος της συζήτησης. Ζητάμε σταδιακή κατάργηση όλων των, χρυσών βίζων και λυπούμεθα για το ότι αρκετά κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει κάτι τέτοιο εγκαίρος. Ζητάμε από την Κομισιόν να αξιολογήσει την δυνατότητα σύστασης ενός τέτοιου μηχανισμού είτε ως κάτι το καινούριο ή ως ένα σε ένα εφιστάμενο θεσμικό όργανο. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα των όσων έχουμε επιτύχει. Και τώρα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη πέτυχε πολλά τα τελευταία πέντε χρόνια στην ε, καταπολέμηση της φορολογικής απάτης ε, και του οικονομικού εγκλήματος, αλλά έχουμε και πολλά να κάνουμε. Κάποιες αρχές ε, κρατών μελών δεν έχουν ανταποκριθεί στις ευθύνες τους να συνεργαστούν, να εποπτεύσουν και να τράσουν Κάποιες ε, τράπεζες ε, δεν έχουν ακόμα εκπληρώσει τις ε, νομικές απαιτήσεις για τις βασικές απαιτήσεις για να γνωρίζουν τους πελάτες τους. Και βεβαίως κάποιοι έχουν αποδειχθεί τελείως ανεπαρκή στην ανείχνευση και δίωξη αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων. Αυτή είναι μια σκληρή κρίση στην οποία δυστυχώς καταλήγουμε. Οπότε τώρα λίγα πρακτικά λόγια. Υπάρχει όπως ε, ξέρετε ένα όριο λέξεων των εκθέσεων και αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να προσθέσουμε ε, πέντε σελίδες ε, κειμένου τις οποίες θα καταθέσουμε ως τροπολογίες ε, των εισηγητών και θα καλύπτουν όλες τις θεματικές πτυχές της έκθεσης αυτής. Και αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ξέρετε, δεν έχει τελειώσει ακόμα η δουλειά της Επιτροπής μας. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακροάσεις και επισκέψεις και αυτά βέβαια θα φανούν στην έκθεσή μας και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μέχρι την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Όλα αυτά θα προσθεθούν οπωσδήποτε στις ε, τροπολογίες των συναδέλφων και των πολιτικών ομάδων και έχουμε και κάποιες περιπτώσεις που νομίζω αξίζουν ειδική ε, προσοχής. Να αναφέρω κάποια παραδείγματα λοιπόν. Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλά να κάνουμε για την αποτελεσματική προστασία των καταγγελόντων στην Ευρώπη. Η ακρόαση της προηγούμενης εβδομάδας με τον κύριο Χάουαρτ Μπούγκενσον της τράπεζας Dendenske Bank και των δικηγόρων του νομίζω μας έδειξε το ότι δεν προστατεύονται επαρκώς ε, οι καταγγέλλοντες στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο και στα κράτη-μέλη και στο επίπεδο της Ένωσης ε, και αυτήν την στιγμή έχουμε μια έκθεση η οποία θα αποτελέσει ορόσημο στον τομέα αυτών. Όμως πρέπει να ακούσουμε και τις σύμβουλες ε, που, που μας ε, δόθηκαν για να υπάρξει ειδική νομοθεσία για το θέμα αυτό. Επιπλέον πρέπει να δούμε την χρήση των ε, συμφωνιών εμπιστευτικότητας που γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται για να σιωπήσουν οι ε, δυνητικοί καταγγέλτες, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Επίσης έχουμε δουλειά που πρέπει να γίνει στους φακέλους CUM-X. Οι χειρότερες περιπτώσεις ίσως ε, φορολογικής απάτης που έχουμε δει λόγω του ότι ε, πρόκειται περί καθαρής κλοπής χρημάτων των φορολογουμένων που υποτίθεται ότι θα πήγαινε σε σχολεία, νοσοκομεία κτλ. Τα οποία έκλεψε μια μικρή ελίτ τραπεζιτών για να κάνουν μεγάλη ζωή σε Ντουμπάι και Ελβετία. Αυτό κατέστη δυνατόν λόγω της συγκλονιστικής έλλειψης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Εν ολίγης, οι δράστες ε, του εγκλήματος αυτού έκαναν ε, όλα αυτά που δεν είχαν κάνει τα κράτη-μέλη. Συνεργάστηκαν, μοιράστηκαν πληροφορίες και εργάστηκαν συστηματικά για να επιτύχουν τους στόχους τους. Εμείς ως αρμόδια επιτροπή πρέπει να εξηχνιάσουμε αυτό το σκάνδαλο ε, για να φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, αναμένω την συζήτησή μας και την συνεργασία μας έχοντας ε, συνεργαστεί σε όλες τις ειδικέ επιτροπές και έχοντας ε, την τιμή να έχω υπάρξει εισηγητής να κάνω μια τελευταία παρατήρηση. Η εργασία μου στην Επιτροπή αυτή νομίζω συνομαδευτική από ένα μεγάλο βαθμό συνεργασίας και ακαιρεότητας ε, και εργαστήκαμε νομίζω σε ένα πολύ σωστό πνεύμα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους και αναμένω μια επικοδομητική συνεργασία μέχρι το τέλος της ε, θητείας μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ θερμά τους δύο συνεισηγητές για την εργασία τους. Νομίζω ότι είναι πολύ αντικειμενική έκθεση που καθιστά σαφές ότι εργάστηκε πολύ η Επιτροπή, έκανε πολλές έρευνες. Εκεί όμως που δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος είναι το θέμα των συγκεκριμένων προτάσεων. Σε τελευταία ανάλυση, αν θέλουμε να έχουμε κάποια επίδραση, πρέπει να κάνουμε εντελώς συγκεκριμένες προτάσεις για το τι πρέπει να αλλάξει. Και να μην ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για απίστευτα ποσά. Αν επιτύχουμε ακόμη και ένα σημαντικό τμήμα αυτής της φοροδιαφυγής να το αντιμετωπίσουμε, να το ε, καταργήσουμε δηλαδή, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να καλύψουμε το επόμενο πολιτέ πλαίσιο. Δεν θα καθόλου, καθόμαστε καθόλου να συζητάμε για το 1,1 ή το 1,3 του ΑΕΠ. Είναι σαφές ότι η βελτιστοποίηση της φορολόγησης έτσι όπως αποκαλείται είναι απαράδεκτη. Το θέμα είναι αν κάνουμε ε, τα σωστά βήματα. Η φοροαποφυγή για παράδειγμα. Και ακούω να ε, φορολογήσουμε τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών για να υπάρξει έτσι κοινωνική δικαιοσύνη. Νομίζω ότι στην ουσία παραπλανόμεθα. Τα στοιχεία που αναφέρονται είναι μία προσωμείωση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτοί οι οποίοι πρώτοι πρότειναν αυτά τα στοιχεία είπαν ότι δεν χρησιμοποιούνται σωστά και τα απέσυραν. Και είπαν ότι δεν πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία αυτά σε σχέση με το όνομά του. Είναι λάθο στοιχεία. Αυτό που πληρώνει μια ψηφιακή επιχείρηση σε σχέση με αυτό που πληρώνει μια κανονική εντό αγωγικών επιχείρηση δεν διαφέρουν πολύ. Πολύ λιγότερο από ό,τι ε, παρουσιάζεται. θα πρέπει κυρίως να στραφούμε προς τη φορολόγηση του κύκλου εργασιών. Υπάρχουν τρεις τομεί όπου υπάρχουν ε, άσχημες καταστάσεις. Πρώτα απ' όλα ο ΦΠΑ. Εδώ και 40 χρόνια συζητάμε για τι απάτες του ΦΠΑ. Ξέρουμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν το κάνουμε. Εδώ τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Και πολύ σοβαρότερα. κάνουν διάφορε αναλύσεις και μελέτες και τίποτα άλλο. Ιδίω το κουμ και το κουμ και αυτό το NDA που προέκυψε πριν από δύο εβδομάδε. δεν είναι δυνατόν να ε, είναι αρμόδιες οι εθνικές ε, φορολογικές αρχές μόνο για τη φορολόγηση και όχι για την εποπτεία. Χρειαζόμαστε οι τράπεζες που έχουν διεθνή παρουσία να υπογράψουν μία υπεύθυνη δήλωση δεσμευτική ότι δεν θα στηρίζουν τέτοιου τύπου συναλλαγέ. Αλλιώ αυτό θα είχε συνέπειε. Θα του στέλναμε τον εισαγγελέα. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, για τους ε, λογιστές, τους ελεύθερους επαγγελματίε που στηρίζουν τέτοιες ε, ε, καταστάσεις να απογορευτεί η άσκηση επαγγέλματος διαβίου θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα είδος ε, ευρωπαϊκού FBI και να έχουμε έντονη συνεργασία με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί όπως μας εξήγησαν χθες ε, κάποιοι ειδικοί, αυτό δεν είναι πλέον δυνατόν, στην, τέτοιου τύπου απάντες δεν είναι δυνατόν να διεξαχθούν στην Αμερική. Οι καταγγέλλοντες βεβαίω πρέπει να προστατεύουν, αλλά όχι μόνοι αυτοί. Μόνον αυτοί. Ακόμη και οι δημοσιογράφοι που κάνουν έρευνες, αντιμετωπίζουν δυσχέρειες οι οποίοι ε, διώκονται από δισεκατομμυριούχους και δεν είναι σε θέση να πληρώσουν 200-300 ε, ευρώ δικαστικά έξοδα για να ε, ε, ε, τον εαυτό τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μικέλ Ουρμπάν Κρέσπο, 4 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρο, θα, Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου. Η δομή της ε, έκθεσης ε, είναι καλή, πιστεύουμε. Είναι καλές οι μέθοδοι εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό που μας ανησυχεί ωστόσο είναι ότι οι συγητές ε, λένε ότι μην είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν το περιεχόμενο της έκθεσης με άλλες πολιτικές ομάδες. Γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές δημιουργείται μια δυναμική ευρείας ε, πλειοψηφία που δεν έχει τελικά αποτελέσματα. Θα ήταν καλύτερα να είχαμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις των σχεδόν προηγουμένως. Αυτή η η λογική ευρεία πλειοψηφία και αποκλεισμού κάποιων άλλων που είχε ω αποτέλεσμα να μην λάβουμε εμεί θέση αντιπροέδρου, ελπίζουμε να μην διατηρηθεί στι διαπραγματεύσει για την τελική έκθεση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κάτι που είναι θεμελιώδες για μας είναι ότι η πραγματικότητα είναι πολύ ε, βαριά, ε, απογοητευτική. Διαπιστώνουμε ότι τρέχουμε από πίσω. Είμαστε τελευταίοι και καταϊδρωμένοι. Η πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν καταφέραμε να λύσουμε τα αντιδραστοτικά προβλήματα που κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση έφορο έδαφος για τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Για παράδειγμα, η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, κεφαλαίων, το τραπεζικό απόρριτο, η ύπαρξη φορολογικών παραδείσων και εντό τη Ένωση και στην περιφέρειά τη. Είναι ταμπού αυτά τα θέματα, δεν τα συζητάμε. Αλλά είναι όπω ε, στην πισίνα, ξέρετε τα πράγματα. Αν υπάρχει κάποιο, κάπου στα ατυχώματα τη ε, πισίνα. Μία ε, μικρή ε, σχισμή φεύγει από όλο το νερό και μας δεν είναι μικρή σχισμή, είναι τρεπιτήρι. Θέματα τα οποία τα έχουμε εγκρίνει σε προηγούμενες εκθέσεις. Στο ΠΑΝΑ, στο ΤΑΞ 1, στο ΤΑΞ 2. Εγκρίναμε κι εμείς και ως ολομέλεια ε, συστάσεις. Δεν περιέχονται σε αυτή την ε, πρόταση έκθεσης. Η τάξη 3 λοιπόν ε, υπολείπεται ε, ε, των αποφάσεων που έχει λάβει προηγουμένως το Κοινοβούλιο. Τι υποχωρήσει έχουν γίνει, για παράδειγμα. Γιατί μιλάμε για ενδιαμέσους και όχι διευκολυντές. Δεν είναι σωστό αυτό. Η έκθεση πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο τμήμα για αυτούς που διευκολύνουν. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για τις τράπεζες όταν μιλάμε για το ξέπλυμα χρήματος. Διότι τα διάφορα σκάνδαλα ε, αποδεικνύουν ότι συμμετέχουν παντού σε κάθε είδους ε, απάτες. Η έκθεση Πάνα ήταν πολύ πιο σαφής. Για παράδειγμα, πώς πρέπει να τιμωρούνται αυτοί που διευκολύνουν αυτές τις ε, συναλλαγές. Και το κομμάτι για τις φορολογικές αμνηστίες που δεν καταδικάζονται, ενώ η Πάνα το καταδίκαζε, η έκθεση της Επιτροπής Πάνα. Βλέπουμε λοιπόν οι παναχωρήσει σε σχέση με προηγούμενες εκθέσεις. και για τι επιχειρήσει βιτρίνα. Δεν αρκεί η έκθεση να λέει ότι ότι ε, δεν έχουν επαρκή οικονομική δραστηριότητα σε χώρες όπως η Κύπρος, το Λουξεμβούργο. Πρέπει να λέμε ότι αυτό είναι σαφής ένδειξη φορολογικής ε, φοροδιαφυγής. Η έκθεση Πάνα ήταν πολύ πιο σαφής από όλων αυτών. Επίσης η έκθεση Πάνα ήταν πολύ πιο σαφής για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ε, συνεργασίας για την καταπολέμηση των ε, απατών. Πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση. Και η ίντα επίσης είχε κάνει μια έκθεση το 2016 για αυτό το θέμα που θα, μπορούσατε να, θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που αναφέρονται αλλά θα έπρεπε να είναι πολύ πιο επικριτικά. Για παράδειγμα, ο κατάλογος των φορολογικών παραδείσων είναι αστείο. Δεν αναγνωρίζει κανένα φορολογικό παράδεισο εντό τη Ένωση, αλλά ε, αναφέρει μόνο έξι χώρε που είναι όλε ε, αναπτυσσόμενε. Κατά λίγο. Επίση. Το BEPS είναι ανεπαρκές. Θα πρέπει να στηρίξουμε μία ενιαία παγκόσμια φορολόγηση και να γίνει ε, αναδιαπραγμάτευση κάποιων φορολογικών συμφωνιών που να, ούτως ώστε να καταλήξουμε ε, να, καταλάβουμε, σωστά πώς λειτουργούν οι πολυεθνικές. Αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια των Ηνωμένων, των ε, και όχι του ΟΣΑ. Πρέπει να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα, διότι σε μισή ώρα καταφθάνει ο Επίτροπος. Σβέν Γκίγκολντ για τους Πρασίνους για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχάς τους συνεισηγητές για το σχέδιο κειμένου. Δεν είδα μέχρι τώρα να υπάρχει μία προσέγγιση και συμμαχία όσον αφορά την οτροπία ε, κατ' παρελθόν και δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ε, ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία πέρα από πολιτικό τοπίο, ε, πέρα από τις πολιτικές συμμαχίες. Στην έκθεση περιέχονται διάφορα καλά σημεία και είναι σημαντικό να κάνουμε σύγκριση των επιτευμάτων των προηγουμένων επιτροπών, να μην λησμονούμε κάποιες από τις σημαντικές εκκλήσεις που είχαμε απευθύνει κατά το παρελθόν, ακόμα και αν αυτά δεν εφαρμόστηκαν, και να σημειώσουμε και τα όσα έχουν εφαρμοστεί. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε πολύ σαφέστερη διατύπωση να φαίνεται ότι κάποιες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα έχουν κολλήσει στο Συμβούλιο, όπως η υποβολή εκθέσεων αναχώρα και η κοινή ενοποιημένη βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Αυτά είναι στοιχεία που αποτελούν τη ρίζα των προβλημάτων και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να πιέσει τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε εκείνα να επιφέρουν τι αναγκαίε νομοθετικέ αλλαγέ. Πρέπει να εκφραζόμαστε ανοιχτά για την έλλειψη συνεργασία από πλευρά Συμβουλίου, που δεν μοιράζεται μαζί μα έγγραφα. Και η Βουλγαρική Προεδρία επανειλημμένα αρνήθηκε να έρθει στην Επιτροπή. Αυτό αποτελεί παραβίαση της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας. Και θα πρέπει να αποφύγουμε να το πούμε σαφώς. Όσον αφορά την φορολόγηση επιχειρήσεων, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην οδηγία DAC 3 όσον αφορά τα tax rulings και σε κάποια τμήματα της ως επιχειρήσεων έχουμε μειοδοτική τάση, κυρίως όσον αφορά τα θέματα ευρεσιτεχνίας και τα, το, τους φορολογικούς συντελεστές. Θα πρέπει να εκφραζόμαστε ανοιχτά επίσης για τη διάδοση ε, της μειοδοσίας ε, όσον αφορά ε, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Πολλούν κάποια κράτη-μέλη διαβατήρια που επιτρέπουν να μετακινήσεις την, τον τόπο διαμονή σου και να πας σε ένα κράτος μέλος όπου έχεις πιο ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση και επιτρέπουν ε, σε πλουσίου ειδικό φορολογικό καθεστώ σε κάποιε χώρε όπω είναι η Ιταλία. Αυτό είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εδώ η Ευρώπη όπω κάναμε και με, ε, με τη φορολόγηση επιχειρήσεων. Υπάρχουν μεγάλα κενά στην οδηγία για διοικητική συνεργασία που είχαμε υπερψηφίσει. Το εισόδημα Φερρυπίν που προέρχεται από στοιχεία ενεργητικό όπως είναι η ιδιοκτησία δεν συμπεριλαμβάνεται και στο ξέπλυμα χρήματο είχαμε διαπιστώσει το ίδιο όπω και με τη φορολογία. Σε κάποιου τομεί κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στην καθημερινή ζωή όσον αφορά το μίστομα και ε, δεν υπάρχει αναγκαία συνεργασία όσον αφορά τι πληροφορίε σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να υπάρχει κανονισμό για τα κρυπτονομίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το συζητήσαμε επανειλημμένα εδώ θεωρούμε ότι πρέπει να εκφραστούμε για τις αρνητικές συνέπειες που υπάρχουν για τις αναπτυσσόμενες χώρες, εκεί που να τα καταφέρουμε καλύτερα. Και τέλος θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή διατύπωση για διάφορες πτυχέ της νομοθεσίας. Και τέλος, από το σκάνδαλο COMEX θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ε, ομοσπονδιακή αστυνομία FBI ή οικονομική αστυνομία για να μπορεί να ε, προστατεύει τους πολίτες μας κατά του οικονομικού εγκλήματος. Διότι το διεθνές έγκλημα κινείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άρα χρειάζονται ευρωπαϊκοί φορείς που θα μπορούν να ε, καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο το διεθνές. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους εισηγητές, εισηγητές. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ένα δεύτερο γύρο. Ο Τόμ Βαντέκελάρ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω και εγώ τους ε, συγητές. Είναι μια πληρέστατη έκθεση και επιπλέον η έκθεση ξεκινάει από γεγονότα και δεδομένα. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά των εισηγητών αλλά θεωρώ ότι κάνει έτσι απλούστερη την συζήτηση και θα ωφελήσει την αξιοπιστία της ε, Επιτροπής μας. Λοιπόν, και αυτό μπορεί να κάμψει και τυχόν αντιρρήσεις. Κάποια πράγματα τώρα για την απάτη του ΦΠΑ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πόσο διαδεδομένο είναι το φαινόμενο και τι θα γίνει με τον εξυγχρονισμό του στήματος ε, ΦΠΑ. Έχουμε λοιπόν αυτό το κενό του ΦΠΑ το οποίο για το Βέλγιο υπολογίζεται σε 3,1 δισεκατομμύρια ενώ γνωρίζουμε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2019 ήταν 2,1 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε έναν ίσως κελισμένο προϋπολογισμό. Θεωρώ ε, κρίσιμο το ότι πρέπει να γίνουν η παραδειγμα παραδείγματο χάρη στο θέμα του ΦΠΑ εκεί πέρα πρέπει να αναλυθεί ευρωπαϊκή δράση. Να δούμε δηλαδή τους κανόνες για το ενδοκινοτικό εμπόριο και τις ε, σχετικές ε, παράνομες ε, κατασκευές. Δεύτερον, οι χρυσές βίζες και εδώ πέρα πρέπει να είμαστε κάπως πιο εντονοί στην επικοινωνία μας αλλά και στο κείμενό μας υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος ε, ξεπλήματος ε, χρήματος ε, και έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες μας. Τέλος, για τα κρυπτονομίσματα, εδώ πέρα ζητάμε ακριβώς η Κομισιόν να κρίνει την κατάσταση και να υποβάλει κάποιες αποτελεσματικές προτάσεις έτσι ώστε πρώτον να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να προστατευτούν οι επενδυτές και να υπάρχει δυνατότητα ε, οικονομικής καινοτομίας και δεύτερον να προλάβουμε τις ε, περιπτώσεις ε, φοροδιαφυγής. Γενικά είμαστε πάρα πολύ θετικοί απέναντι στην έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ σας η Alice Line έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές για τη δουλειά που έκαναν και το ψήφισμα στο σύνολό του είναι αρκετά προχωρημένο. Τα μέλη αυτής της Επιτροπής έχουν αναπτύξει τεχνογνωσία επί φορολογικών θεμάτων και αυτό αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα του κειμένου. Το ψήφισμα χρειάζεται κάποια ενίσχυση σε κάποια σημεία όσον αφορά τις εξελίξεις στα φορολογικά θέματα. Το θέμα των φόρων πρέπει να εξεταστεί και πώς το ΦΠΑ επηρεάζει την ανάπτυξη των αντισωμένων χωρών. Ο φόρος ε, στο ΦΠΑ, το ΦΠΑ είναι από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τη συλλογή πόρων από τις κυβερνήσεις. Πρέπει να καταπολεμήσουμε όμως και την ε, Θέλουμε προοδευτική φορολόγηση να προωθήσουμε κυρίως αυτές τις χώρες. Διότι δεν θέλουμε φαύλο κύκλο περικοπών πόρων για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και για την πρόνοια. Και χρειαζό... Όταν ψηφίσαμε ένα ψήφισμα το 2015 για το πώς θα βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να καταπολεμήσουν φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, χρησιμοποιήσαμε τη λέξη διακυβερνητική, διότι θα πρέπει ε, να μην αποδυναμώνουμε το κείμενο όσον αφορά αυτό το θέμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν αυτό που ζητούσαμε σε εκείνο το ψήφισμα. Δηλαδή ανάλυση ε, των συνεπιών που έχει η ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική και η πολιτική φορολογική των Κατών μελών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μόνο ότι το τρόπος μπορούμε να εντοπίσουμε και να αποφύγουμε επιβλαβεί συνέπειε για αυτές τις χώρες. Γι' αυτό θα προτείνω να προσθεθεί με τέτοια αναφορά στο κείμενο. Πέραν αυτού, η κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών πρέπει να ανακατανεμηθεί και να βασιστούμε στο καλό παράδειγμα ε, της συμβάσεως για τη φορολόγηση του ΟΗΕ. Ήταν πολύτιμο στοιχείο που μάθαμε από τις ε, δημόσια κράσεις μας και κάποιες τολμηρές τροπολογίες ε, ε, θα αναφέρω όσον αφορά τη διαπραγμάτευση φορολογικών συνθήκων από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αν μιλήσουμε μια φωνή, θα είναι κάτι αποτελεσματικό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι κάτι και πιο δίκαιο για τι χώρε εταίρου. Ελπίζω η συνεισφορά μου να ενισχύει έτσι περαιτέρω αυτή την έξοχη έκθεση. Ευχαριστώ. Ο Βολφ Κλίντ για την Άλντε. Ίσως σε αυτή τη χρονοθυρίδα να μιλήσω εγώ να κάνω ένα σχόλιο, όχι επί της ουσίας τόσο, αλλά επί της προσεγγίσεως. Να επενθυμίσω κάτι. Δεν είναι μια συνηθισμένη έκθεση επιτροπής. Δημιουργήθηκε, συστήθηκε αυτή η επιτροπή για την εκπόνηση μιας εκθέσεως. Θα γίνουν διάφορες αποστολές, ακροάσεις, ε, έγιναν προσπάθειες. Ε, αυτό κόστισε αυτό είναι ένα θέμα που θα θίξω. Η έκθεση πρέπει να υπογραμμίζει το έργο και των τεσσάρων επιτροπών σε αυτόν τον τομέα. Ε, έργο που επιτελέσει κατά τη θητείας. Από την αρχή της θητείας μας είχαμε πει ότι πρέπει να εστιαστούμε επί αποτελεσματικής εφαρμογής και να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος των συστάσεων προηγουμένων επιτροπών. Εν γέννη αυτή η έκθεση πρέπει να είναι η Rolls Royce των εκθέσεων. Πρέπει να είμαστε σαφείς ποια είναι η μορφή της υλοποίησης των συστάσεων. Πρέπει να είμαστε σαφέστατοι όσον αφορά νέα πορίσματα και νέες συστάσεις. Αυτά τα σχόλια είχα. Σφεν Γκίγκολτ για τους Πασίνους έχει το λόγο. Και αν έχουμε άλλους θα χρειαστεί. Όχι. Μ' ακούσατε πολύ σε αυτή την επιτροπή και αρκεί για σήμερα, λέει και ο Κίκολτ. Άρα, φαίνεται ότι ήμασταν αποτελεσματικότατοι στις εργασίες μας. Οπότε η διαδικασία κάτσε διά ξεκινά. Ο Πολ Τάγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές. Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ επικοδομητική έκθεση. Εν συντομία, θα να πω κάποια πράγματα. Πολύ δύσκολο το θέμα της ελλείψεως στοιχείων και η δυσκολία αναλύσεως των διαθεσίμων στοιχείων. Καμιά φορά δουλεύουμε στα σκοτεινά. Αυτό πρέπει να το αναφέρει η έκθεση. Χρειάζεται ερευνητική υποδομή στην Ευρώπη. Διαθέσιμα στοιχεία να τα διαθέτουν οι εθνικές φορολογικές αρχές. Να βελτιωθεί και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για αυτά τα θέματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το πρώτο. Ε, ένα παράδειγμα είναι ο φόρο για τις ψηφιακές υπηρεσίες που συζητούμε αυτέ τις εβδομάδες. Δεύτερο, κάτι που λείπει από την έκθεση. Η επαφή μεταξύ κατών μελών παραμελείται η συνεργασία τους και η διάδραση. Υπάρχουν σημαντικές ροές μεταξύ κρατών μελών εις βάρος των χωρών που έχουν υψηλότερο συντελεστή φορολογικό και η ροή είναι προς τις χώρες με χαμηλότερο συντελεστή. Είμαι από την Ολλανδία και μπορώ να πω ότι πολλά από τα χρήματα πάνε από τη Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία πάνε στην Ολλανδία και πρέπει ε, να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θα πρέπει ένα κράτος μέλος να κινείται εις βάρος των άλλων κρατών μελών. Άρα χρειάζεται ευρωπαϊκή προσέγγιση. Το υποστηρίζει αυτό το κοινοβούλιο όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Αντί κεντρική αντιμετώπιση του ξεπλήματος χρήματος, να βρούμε άλλη διατύπωση. Ε, παραδείγματος χρειάζεται και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδιακή Αστυνομία, ένα Ευρωπαϊκό FBI. Άμα έχουμε διασυνοριακό έγκλημα, χρειάζεται και διασυνοριακή δίωξη. Πρέπει να βρούμε μια λύση όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρειάζεται και στήριξη και του λαού πάνω σε αυτό για να το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Πύρκου Ευχαριστώ πολύ. Τους συναδέλφους ε, που συνεργάστηκαν για την εκπόνηση αυτού του κειμένου και τη γραμματεία που τους βοήθησε. Η Επιτροπή αυτή και οι προηγούμενες έχουν εργαστεί σκληρά για να αντιμετωπίσουν την, οργανωμένη, την οργανωμένη εγκληματικότητα. Υπάρχουν επίσης και δημοσιογράφοι ε, που κάνουν έρευνες ε, καθώς και καταγγέλλοντες οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει για παράδειγμα στην περίπτωση του Κούμεξ, του σκανδάλου Κούμεξ. Θέλω να ασχοληθώ ιδιαίτερα με το θέμα των χρυσών βυζών. Δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, δημιουργούν κινδύνους ε, ακόμη και από πλευράς ασφαλείας. Και αυτό αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Ακόμη και τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν τέτοιους, ε, τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι δυνατόν ε, να πληρώνει κανείς και γίνεται πολίτη της Ένωσης. Σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το πόσε αιτήσει έχουν υποβληθεί, πόσε τέτοιε βίζε έχουν χορηγηθεί κτλ. Μ' αρέσει η εξέλιξη της έκθεση, η κατεύθυνση τη δηλαδή. Ελπίζω λοιπόν να καταργήσουμε τέτοιου κανόνε για χρυσέ βίζες και παρακολουθώ και την έρευνα που κάνει η Κομισιόν και τις συστάσεις που κάνει για το θέμα αυτό στο μέλλον. οι υπάλληλοι μα θα πρέπει να επιδεικνύουν και περισσότερη πρωτοβουλία όταν γίνονται τέτοιε αποκαλύψει. Μόλις ε, γίνονται γνωστές τέτοιες καταστάσεις, θα πρέπει οι υπηρεσίε και οι υπάλληλοι να αναλαμβάνουν το ρόλο το, να παίζουν και το ρόλο του μετά που τα έχουν αποκαλύψει δημοσιογραφικά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο. Ο Βολφ Κλίντ. νομίζω ότι η τάξη μεγέθους ε, των φοραπατών που συζητάμε είναι γνωστή στη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού. Γιατί τα λένε τα μέσα. Τα γράφουν. Κατά τη γνώμη μου. Η κοινή γνώμη θεωρωτάται. Μπορώ να έχω καμιά εμπιστοσύνη στην Ένωση να τη θεωρώ δηλαδή ένωση δικαίου και αν αυξάνονται οι αμφιβολίες θα αρχίσουν ε, να αμφιβάλλουν ε, και για το εάν και κατά πόσο η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Δεν πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ελαφρά. Δεν είναι θέμα απλώς να βρούμε τα κλεμμένα που έχουν κλέψει οι εγκληματίες από τους φορολογούμενους. Αν δεν βρούμε μια λύση, υπάρχει κίνδυνος ε, υπονόμευσης των θεμελίων της ε, Ένωσης και της δημοκρατία μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στις συστάσεις μας για να αποδείξουμε στους πολίτες, τώρα που επίκυνται οι ευρωεκλογέ, ότι όντως προσπαθούμε να τους πιάσουμε. Γιατί όταν τους πλησιάζουμε αυτοί πατάνε γκάζι και εξαφανίζονται. Σκληρός αγώνα, αλλά αν δεν κερδίσουμε θα χάσουμε. Πολλά. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρο. Δεν βλέπω να θέλει κανεί άλλο το λόγο. Οπότε να ευχαριστήσω και εγώ τους συνεισηγητές για τη μέχρι του εργασία τους και τους δίνω το λόγο για τις ε, καταληκτικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα ο κύριος ε, Νίντερ Μακ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να συμπεριλάβουμε και τα πορίσματα των ακροάσεων που είναι εν εξελίξη. Αυτά για παράδειγμα που αποκαλύφθηκαν χθες στη συζήτηση για το ΚΑΜΕΞ. Καλώς ορίζω την έκκληση που γίνεται για πιο συγκεκριμένες ειδικέ συστάσεις και βεβαίως ε, με χαρά θα δω τις τροπολογίες σας τις οποίες και θα συζητήσουμε. Δεν είναι η πρόθεσή μας να είμαστε ακριβείς και ειδικοί αλλά ορισμένες φορές ε, δεν είναι εύκολο να βρεις ακριβώς τη λύση. Νομίζω ότι δεν αρκεί η δημιουργία νέων θεσμών για να επιλύσουμε τα παλιά προβλήματα αλλά να δω τις συστάσεις σας βεβαίως. Και τέλος, Προφανώ μα ενδιαφέρουν και οι συστάσει που έχουν γίνει σε προηγούμενα κείμενα του Κοινοβουλίου και καταλαβαίνουμε ότι κάποιε προτάσει, όπω οι προτάση για το CCCTB μπορούν να λύσουν πολλά προβλήματα στον τομέα τη φορολόγηση. Ελπίζω λοιπόν να αναφερθεί στι τροπολογίε. και επίση ευχαριστώ τον Μπολ ιδιαίτερα που ανέφερε το πρόβλημα ε, ελλειπών στοιχείων. Στην έκθεσή μα, προσπαθούμε να βασιστούμε όσο είναι δυνατό σε στοιχεία, σε γεγονότα. Αλλά αν έχουμε καλύτερα στοιχεία, θα έχουμε και καλύτερα πορίσματα και καλύτερες συστάσει. Θεμελιώδε αυτό λοιπόν. Βεβαίω, προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία για να επιτύχουμε συμβαστικές τροπολογίες. Πολλέ καλέ ιδέε μπορούμε ακόμη να συμπεριλάβουμε στην έκθεση και θα εργαστούμε με όλες τις ομάδες για να βρούμε ε, τους καλύτερους δυνατούς συμβασμούς. Ο κύριος Κόφοντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους συναδέλφους. Πολύ επικοδομητικά αυτά που μας είπαν. Στον κύριο Κλίντς, έχετε απόλυτο δίκιο στην τελευταία παρατήρησή σας. Η εφαρμογή, η αυστηρή εφαρμογή ε, της νομοθεσίας είναι θεμελιώδες θέμα. Και στα θέματα φορολόγησης και οικονομικού εγκλήματος ε, προφανώς δεν εφαρμόζεται παρκώς ο νόμος από τα κράτη-μέλη, από τις διάφορες υπηρεσίε. Πρέπει λοιπόν να προτείνουμε λύσεις για να καλυφθεί αυτό το κενό. Τώρα το μήκος της έκθεσης, ξέρετε, επαναλαμβάνω, υπάρχει όριο. Θα είχαμε συμπεριλάβει πολλά άλλα θέματα στην έκθεση αλλά δεν γινόταν. Έπρεπε λοιπόν να θέσουμε προτεραιότητες. Και οι εκθέσει των άλλων επιτροπών, τάξ 1, τάξ 2 πάνω, οι συστάσει του και οι κλήσει που κάνουν ε, για περαιτέρω ενέργειες εξακολουθούν να ισχύουν. Είναι πολιτική του Κοινοβουλίου. Αν έπρεπε να τα επαναλάβουμε όλα αυτά, δεν θα υπήρχε χώρο για να προσθέσουμε τίποτα καινούριο. Υπάρχει περιορισμός ε, του αριθμού σελίδων. Βασιστήκαμε, όπω είπε και ο πρόεδρο σωστά, στην εργασία όλων των συναφών τεσσάρων επιτροπών. Και συμφωνώ με τον κύριο Γκίγκολτ, ιδιαίτερα για το CCCTB και για τι αναχώρασει τάσει και εκθέσει. Πρέπει να το τονίσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για τα θέματα αυτά πριν το τέλο τη θητεία. Πρέπει να κάνουμε έκκληση ω Επιτροπή να καλέσουμε κράτη-μέλη να προωθήσουν τα θέματα αυτά. Και για την ειλικρινή συνεργασία. Τονίζουμε ότι δεν θεωρούμε ότι το Συμβούλιο συνεργάζεται τόσο ειλικρινώς όπως ε, ε, καθορίζουν οι συνθήκες. Θα το βάλουμε αυτό. Αυτές οι ειδικέ επιτροπές δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους αν δεν έχουν πρόσβαση στην αναγκαία πληροφόρηση και τα στοιχεία που ε, διαθέτει το Συμβούλιο. Τώρα να μην πω σε άλλες λεπτομέρειες, σημείωσαμε τα σχόλια. Άλλοι ανέφεραν ότι μετά τα έγγραφα του Παραδείσου έχουμε συμπεριλάβει και άλλα θέματα και συγκεκριμένα την καταπολέμηση του, της απάτης ε, επί του ΦΠΑ για παράδειγμα για, με τα γιότ, με τα ιδιωτικά αεροπλάνα αλλά είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα Κυρία Σλάιν Κοιτάξτε, λέτε ότι αναφέρουμε αναπτυσσόμενες χώρες. Η εργασία μας πρέπει πάντα ε, να συνδυάζεται με την αναπτυξιακή πολιτική. Η φορολογική μας πολιτική με την αναπτυξιακή μας πολιτική. Βεβαίως. Πρέπει να είναι συνδυασμένη η πολιτική μας. Θεμελιώδες αυτό. Να υπάρχει συνέπεια δηλαδή μεταξύ των διαφόρων πλευρών της πολιτικής μας. Με τις βασικές ε, αρχές μας. Για την εφαρμογή τώρα. Γιατί έχουμε εγκρίνει πολλά καλά νομοθετήματα. Καλούμε να υπάρξει κατά την επόμενη θητεία μία υποεπιτροπή για θέματα φορολογίας. Γιατί πολλά από τα θέματα αυτά, αυτά που θα προτείνουμε εμείς και αυτά που έχουν ε, εγκριθεί από προηγούμενες επιτροπές, πρέπει να εφαρμοστούν. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει το κατάλληλο όργανο στο Κοινοβούλιο για να ε, καλή και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Στον Πολ τώρα. Συμφωνώ η έλλειψη στοιχείων. Και η... Ε, παρουσίαση χονδρικών στοιχείων, προσεγγιστικών στοιχείων, δεν μας βοηθάει. Χρειαζόμαστε καλύτερα στοιχεία για να έχουμε καλύτερες προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ, προσβλέπω στη συνέχιση της διαδικασίας όχι, όχι, δεν επιδιώκουμε ευρείε πλειοψηφίε. Όχι, Μιγκέλ, Θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα με όλου μαζί για να βελτιώσουμε την έκθεση με βάση τα στοιχεία ε, που έχουμε συλλέξει. Έτσι πρέπει να εργάζεται μια ειδική επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ε, δανούς εκπαιδευόμενους ε, δημοσιογράφους ε, στα θεωρία και ευχαριστώ τους εισηγητές, τους κοιόδης εισηγητές για την δουλειά τους και όλους όσους μίλησαν σήμερα για την πολύ αποτελεσματική αυτή συζήτηση που καταφέραμε να τελειώσουμε και λίγο νωρίτερα Οπότε κάνουμε ένα διάλειμμα ολίγων λεπτών για να ξεκινήσουμε στις 4 με τον Επίτροπο τον κύριο Μοσκόβηση.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

Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνουμε τις εργασίες ε, της Επιτροπής μας. Τάξε 3. Καλώς ορίζοντα θερμά τον Επίτροπο Μοσκοβισή. Πού θα μας μιλήσει για την εφαρμογή των συστάσεων ε, άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου κατά την τρέχουσα θητεία. Θα μας μιλήσει επίσης για το ΕΚΟΦΗΝ του Δεκεμβρίου που θα πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις για την ε, φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Υπάρχει και το θέμα του γκρίζου καταλόγου φορολογικών παραδείσων. Πολλά θέματα έχουμε να συζητήσουμε λοιπόν μαζί του. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επίσκεψή του, για τη δεύτερη επίσκεψή του. Και ευχαριστώ για την καλή του διάθεση και την καλή συνεργασία που έχουμε με το Κοινοβούλιο, που έχει με το Κοινοβούλιο. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Παρακαλώ ε, μία πρώτη παρουσίαση 15 ε, λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, την οποία όπως πάντα χαίρομαι ιδιαίτερα να αποδέχομαι. Εδώ και πάνω από 8 μήνες η Επιτροπή σας ε, εργάζεται και έχει ακόμη 4 μήνες εργασίας μπροστά της. Καλή συγκυρία λοιπόν για να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχουμε σημειώσει στη κοινή πάλι κατά της ε, φοροδιαφυγής και της φοροαπάτης και λέω κοινή πάλι, γιατί πραγματικά η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ε, συνεργάζονται στενά. Οι ειδικέ επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου για τη φορολόγηση στην Ευρώπη και τις φορολογικές πρακτικές, tax, tax 2, πανά, μετά από τα διάφορα, φορολογικά σκάνδαλα, το LuxLeaks, τα έγγραφα του Παναμά, τα, τις διαρρές του ποδοσφαίρου και πιο πρόσφατα το Κουμέξ. Όλα αυτά αποδεικνύουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αποφασιστικότητα ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και επέβαλε ε, ένα ρόλο απαραίτητο στην καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής. Οι δύο θεσμοί μας είναι φυσικοί σύμμαχοι σε αυτόν τον αγώνα και νομίζω ότι έχουμε συνεργαστεί πολύ αποτελεσματικά και σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας, όπως και εσείς πιστεύω ότι βασίζεστε στη δική μου. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συμπολιτών μας. 75% θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για να κατοπολεμήσει την ε, φοροδιαφυγή και τη φοραπάτη. Και θεωρούν ότι είναι προτεραιότητα. Έπρεπε λοιπόν να δράσουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι και τι ευρωεκλογέ, ούτως ώστε το επόμενο κοινοβούλιο και η επόμενη επιτροπή πρέπει να σκεφτόμαστε και τους ε, διαδόχους μας να συνεχίσουν την αποφασιστική προσπάθεια για μια δίκαιη και διαφανή φορολογία στην Ένωση ενώ είμαστε ένα εξάμεινο πριν τι ε, ευρωεκλογέ, πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό τη δράση μα. Νομίζω ότι μπορούμε να είστε περήφανοι για τι προόδου που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια τη ε, τρέχουσα θητεία. Αυτά τα τέσσερα χρόνια γίνανε πολύ περισσότερα από ότι τα προηγούμενα 20. Μαζί αποδείξαμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν καθοριστικές πρόοδοι παρά το, τη δυσχέρεια της ομοφωνίας που στο παρελθόν ε, μας είχε μπλοκάρει. Από το 2014 καταφέραμε να περάσουν με ομοφωνία 13 προτάσει. Αυτό είναι άνευ προηγουμένο. Αυτό δείχνει ότι αλλάζει η νοοτροπία των κρατών μελών. Αυτό δεν έγινε αυτόματα, έγινε κάτω από την πίεση τη κοινή γνώμη, Των σκανδάλων που προέκυψαν. Των διεθνών θεσμών. Και υπό την πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο δείχνει μεγάλη επαγρύπνηση. Οπότε η ε, ε, αδράνεια δεν ήταν πια δυνατή, άλλαξε η ατμόσφαιρα. Κατά τα τέσσερα χρόνια αυτά, δύο αρχές ήταν στη δράση μας και των δύο. Η διαφάνεια και η φορολογική δικαιοσύνη. Για την διαφάνεια, η πιο συμβολική πρόταση είναι αυτή που θέλει να υπάρχει διαφάνεια στην εργασία των ενδιαμέσων, τα δικηγορικά γραφεία, του ε, τους συμβούλους, ε, τις τράπεζες που πουλάνε επιθετικές ε, φορολογικές στρατηγικές. Αλλά πρέπει να υπάρξουν αυστηρότεροι κανόνες σε όλους που κινούνται στα όρια της ε, νομιμότητας. Η οδηγία αυτή θα υποχρεώσει τους ενδιάμεσους ε, για φορολογικά θέματα το 2020 να γνωστοποιούν ε, τα προγράμματα φορολογικής βελτιστοποίησης στις εφορίες. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανένα, αλλά έτσι θα μπορεί ε, η κυβέρνηση να διορθώνει την νομοθεσία αν θεωρεί ότι μειώνει τη φορολογική βάση. Και επίση πρέπει να είναι σαφή η κανόνε του παιχνιδιού των φορολογικών συμβούλων για να αποφευχθούν οι γκρίζε ζώνε. Γιατί κάνεις λιγότερες ε, παράτυπες ενέργειε όταν ξέρει ότι σε παρακολουθούν. Επίσης, γενικεύσαμε την ανταλλαγή πληροφοριών, που είναι η κυριότερη, η μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων. Οι τελευταίες αποκαλύψεις για το θέμα COMEX αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές ελλείψεις και παραθυράκια στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εφοριών, εθνικών εφοριών. Οι ανταλλαγές αυτές ήταν ε, πρώτα απ' όλα εθελούσιες ή με πρωτοβουλία κάποιου. Ε, όλα αυτά έχουν όρια. Αν δεν υπάρχει ε, πραγματική υποχρέωση να υπάρχει η ανταλλαγή πληροφοριών. Από το 2014 λοιπόν προτείναμε να αλλάξουν οι κανόνε του παιχνιδιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αυτές οι ανταλλαγές ε, που στο παρελθόν ήταν ε, ανεπαρκείς, τώρα είναι υποχρεωτικές όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, αποστείλουν σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη όλες τις συμφωνίες για τις τους φόρους που πληρώνουν οι πολυεθνικές, για τις συμφωνίες που έχουν κάνει, το κράτος, που έχουν κάνει τα κράτη με επιχειρήσεις, ούτως ώστε να υπάρχει ισότιμος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη είναι υπέρ ε, του ανταγωνισμού ε, στα φορολογικά. Έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας ε, κάποια κράτη-μέλη. Τα συστήματα αυτά που είναι πλέον εκτικά αξιοποιούνται από κάποιες επιχειρήσεις ή και φορολογουμένους που υιοθετούν επιθετικές φορολογικές ε, στρατηγικέ για να αποφύγουν να πληρώσουν το φόρο που τους αναλογεί. Η... Ο φορολογικός ανταγωνισμός ε, είναι θεμητό, αλλά ο παράτυπος και ακραίο φορολογικός ανταγωνισμός είναι αθέμητο. Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε 7 κράτη-μέλη, των οποίων ε, το φορολογικό σύστημα χρησιμοποιείται πολύ συχνά, κατά τη γνώμη μας, στα πλαίσια της ε, επιθετικής βελτιστοποίησης της φορολόγησης. Ο στόχος μας δεν ήταν να καταδείξουμε κανέναν, να, ε, να εξευτελίσουμε κανέναν. Θέλαμε να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο φορολόγησης που να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης παγκόσμια και ε, ε, έναν ισότιμο ανταγωνισμό. Έχω συζητήσει με διάφορους υπουργούς ε, διαπιστώνω ότι μέχρι και πρόσφατα έχουν υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις. Βέβαια πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη, αλλά λειτουργεί λοιπόν η παρακίνηση και ο διάλογος. Επίσης ε, διεξάγουμε τον αγώνα μας και για τη διαφάνεια και πέρα των ορίων της Ένωσης. Ξέρουμε ότι η φορολογική παράδοση, παράδειση βοηθάνε την φορολογική βελτιστοποίηση. Αναλάβαμε λοιπόν τις ευθύνες μας το Δεκέμβριο του 2017 με δική μας πρότροπη τα, οι 28 Υπουργοί Οικονομικών ενέκριναν για πρώτη φορά έναν κατάλογο των φορολογικών ε, παραδείσων στον κόσμο. Ξέρω ότι ορισμένοι λένε ότι δεν είναι όσε θα έπρεπε να είναι, είναι κάποιοι που δεν έπρεπε και δεν είναι κάποιοι που θα έπρεπε. Αλλά είναι παρόλα αυτά 65 χώρες που καλούνται να λάβουν μέτρα. Και αν δεν τα λάβουν οι χώρες που είναι στον γκρίζο κατάλογο θα περάσουν στον, ε, στο μαύρο κατάλογο, στη μαύρη λίστα. Και πρέπει να ξέρετε ότι είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η τακτική και ορισμένα κράτη που δεν θα τα αναφέρω τώρα έχουν ήδη πάρει μέτρα τα οποία θα μελετήσουμε του χρόνου. Ένα μόνο παράδειγμα. Η Ναμίμπια μετά από τις προσπάθειές της βγήκε από, το, από τη μαύρη λίστα μένουν μόνο 5 ε, από τις 17 χώρε. Σημαίνει ότι πολλοί έκαναν ε, αυτά που έκαναν. Επίσης, θέλω να επιμείνω σε μια πρωτοβουλία φάρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την φορολόγηση της ψηφιακής δραστηριότητας. Γιατί ήταν ε, απόλυτα πιστικό να κάνουμε κάποιες προτάσεις. Γιατί σε λίγα χρόνια μόνο η ψηφιακή δραστηριότητα έχει μετασχηματίσει εντελώς ε, την οικονομία μας και η φορολόγηση δεν ακολουθεί. Πώς να φορολογήσουμε τις ε, φορολογικές δραστηριότητες του ψηφιακού τομέα όταν η φορολόγηση βασίζεται μόνο στη φυσική παρουσία ενώ η δραστηριότητα του ψηφιακού τομέα είναι πολλές φορές άειλε. Είναι επεπαλαιωμένοι οι κανόνες μας. Οπότε τα ψηφιακά κέρδη σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή φορολογούνται πολύ λίγο ή δεν φορολογούνται καθόλου. Αυτό είναι απαράδεκτο έχει γίνει εντελώ απαράδεκτο και στα μάτια των πολιτών μα. Πρέπει να διορθωθεί. Γιατί θα δημιουργούσε και πρόβλημα ε, μακροπρόθεσμα των δημοσιονομικών μας. Έτσι στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Οι ψηφιακές επιχειρήσει και οι επιχειρήσεις των άλλων κλάδων έχουν πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Οι άλλες επιχειρήσεις ε, φορολογούνται κατά μέσο όρο κατά 23% ενώ οι ψηφιακές κατά 9%. Άρα υπάρχει στρέβλωση της φορολόγησης. Έχω υποβάλει δύο προτάσεις στην Επιτροπή για να υπάρχει δίκαιη και ισότιμη φορολόγηση του ψηφιακού τομέα. Η πρώτη, η κυριότερη, είναι εξυγχρονισμός των κανόνων για την εταιρική φορολόγηση εισάγοντα την έννοια της ε, ψηφιακής παρουσίας. Και τη δεύτερη που τη γνωρίζετε είναι αυτή που συζητείτε τώρα και εδώ είναι η ουσία εδώ είναι το ζουμί, το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα πρέπει να αποφασίσει. Έχει να κάνει μία προσωρινή φορολόγηση για, τις, ε, για τα κέρδη ή μάλλον για ε, το φόρο, το κύκλο εργασιών των ψηφιακών δραστηριοτήτων στην Ένωση. Θέλω να τονίσω ότι η στήριξη της πρότασης αυτής έχει διευρυνθεί ιδιαίτερα και θα συνεχίσω να εργάζομαι μέχρι τέλου, ούτω ώστε να υπερβούμε τι ε, αμφιβολίε των κρατών μελών μέχρι το τέλο του έτου. Στι 4 Δεκεμβρίου, ξέρω ότι θα είναι δύσκολο να υπάρξει συνένεση, αλλά δεν είναι αδύνατη. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Αλλά κάτι ευρύτερο, που νομίζω ότι πολλοί θα συμμερίζεστε. Φτάνουμε στα όρια της ε, ομοφωνίας. Ε, λειτουργεί όταν ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε σκάνδαλα, αλλά ε, δεν λειτουργεί όταν πρέπει να κάνουμε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Για ορισμένα πράγματα, ΦΠΑ, CCTV, ενέργεια, ψηφιακό τομέα, ε, έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδο, αλλά δεν καταλήξαμε. Και γι' αυτό αυτή η ομοφωνία. Γι' αυτό θα πρότεινα να παράσουμε στην ειδική πλειοψηφία για τα φορολογικά θέματα από τις αρχές του 2019, όπως ανήγγειλε ο Ζαν Κλοντ Juncker στην ε, ομιλία του για την κατάσταση τη Ένωση. Αν την αποδεχτούν αυτή την ε, μεταρρύθμιση τα κράτη-μέλη, θα αποκτήσουμε πολύ περισσότερο περιθώριο δράση. Θα μπορούμε για αυτά τα βαριά διαρθωτικά θέματα προτεραιότητα που χρειάζονται και αναμένουν οι πολίτε μα να επιτύχουμε περισσότερα. Θα είναι μια πρόοδο τη δημοκρατία. Δεν είναι φυσιολογικό η βούληση ενό και μόνο να υπερισχύει ε, τη όλων των άλλων. Να μην μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα θέλαμε όμω μια ε, έντονη πολιτική στήριξη από το Κοινοβούλιο για να περάσουμε στην ειδική πλειοψηφία. Με το να περάσουμε στην ειδική πλειοψηφία θα περάσουμε και προτάσει για την εσωτερική αγορά και θα διευρύνουμε το πεδίο τη φορολογική πολιτική τη Ευρώπη. Σε αυτό το τομέα δεν έχουμε καθόλου προχωρήσει. Για παράδειγμα, στην προστασία του περιβάλλοντο σε σχέση με αυτό. Ένα φόρο στι ρηπογόνε δραστηριότητε, μια κοινή ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική μέσω τη σωστή και καλύτερα Εναρμονισμένη ενεργειακής φορολόγηση, φορολόγηση τη ενέργειας. Έτσι θα είχαμε και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Πιστεύω ότι, ο, ότι η ομάδα του κώδικα δεοντολογίας μπορεί να επιτύχει πολλά. Είναι δύσκολο οι υπηρεσίε της Κομισιόν να ελέγχουν μόνες τους τους φορολογικούς κανόνες και μέτρα 27-28 χωρών. Αλλά εάν ε, ο κώδικας δοντολογίας που σήμερα δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όπως θα θέλαμε, εάν λοιπόν ε, βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του, πιστεύω ότι θα επιτύχουμε περισσότερα. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα που προσπαθεί να τροποποιήσει τον κώδικα βεντολογίας είναι σύμμαχός μας. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η Ευρώπη έχει ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το τομέα και προασπίζεται ένα πρότυπο ορθής ε, φορολογικής διακυβέρνησης. Ήμασταν οι πρώτοι λοιπόν να υιοθετήσουμε τις δράσεις των ΩΣΑ, ΜΠΕΠΣ. Θυμάμαι σαν υπουργό Οικονομικών ότι αμέσως μετά την Αμερικανική πρόταση και τη γερμανική και βρετανική ε, έγκριση, Ισπανοί, Ιταλοί ε, κλπ. προσήρθησαν στον ΩΣΑ στο πλευρό μας και οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη συμμετείχε ε, στις εργασίες των G20 για την ψηφιακή φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Είχαμε με τρίτες χώρες ε, πρωτοφανή διάλογο. Είμαστε οι πρώτοι ε, με την οδηγία TAD μετά το BEPS χάρη στην πρόθεσή σας και προχωρήσαμε πιο πέρα το ότι η Ευρώπη να γίνει εκπρόσωπος της δίκαιης και σύγχρονης φορολόγησης στον κόσμο και αυτό προσπαθώ να λέω κάθε φορά στο G20 ε, ε, γίνεται σε θα γίνει την Πέμπτη στο Buenos Aires μια συνεδρίαση σε επίπεδο ηγετών των G20. Ε, υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να καταρρευθούμε το χρόνο για να συνεχίσουμε τη μάχη από κοινού. Έξι μήνε απέχουμε από κρίσιμη πολιτική συζήτηση για τα μέσα Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Θα πρέπει να καταδείξουμε την υπεραξία τη ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση και ο φορολογικό τομέα είναι ένα έξοδο τομέα. Είναι ένα θέμα επί το οποίο έχουμε κάνει πολλά ε, και δεν μπορούν να πούν δεν κάνουμε κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτού που φαντάζονται ότι μπορούν μόνοι του να λύσουν το πρόβλημα, νομίζω ότι η ιστορία του έχει διαψεύσει. Ε, απόλυτα. Ε, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκαν, κινήθηκαν σε αυτό το εργοτάξιο από κοινού. Η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να βασιστεί στο επόμενο Κοινοβούλιο, Όπω αυτό ίσχυσε από την αρχή τη θητεία μα. Σα ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα ήταν αποτελεσματικό να δημιουργηθεί μια υποεπιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ε, δεν θα αποφασίσω εγώ. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διοργανωθεί κατάλληλα για το θέμα τη φορολόγηση. Μαζί μπορούμε να οδηγήσουμε σε μια εξέλιξη τη φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο και να γίνει αποτελεσματικότερη φορολόγηση και δικαιότερη. Και εγώ μέχρι τελευταία μέρα θα πολεμήσω ε, για αυτό το σκοπό, μέχρι τελευταία μέρα της παρουσίας μου ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν, ε, ακόμα ένα χρόνο. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Μας αναλύσατε όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ο συνήθως θα έχουμε 5 λεπτά για ερωτήσεις ε, και απαντήσεις. Ένα λεπτό σας ε, παρακαλώ. Ξεκινάμε με τον Λούντεκ Νίντερμαϊερ, ε, τον συνεισηγητή του ΕΛΚ. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ασχολείστε με το θέμα. Έχω τρεις απλές ερωτήσεις. Η πρώτη το Νοέμβριο το 2017 βγάλατε το σχετικό σας έγγραφο για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και μετά κάνετε και τις συστάσεις αναχώρα. Αναρωτιέμαι αν δόθηκε κάποια συνέχεια και αν είχατε κάποια αντίδραση. Δεύτερον, όταν συζητούσαμε την σχετική αμερικανική μεταρρύθμιση εξεφράστηκε η άποψη ότι κόπιες από αυτές τις απόψεις ε, της μεταρρυθμίσης θα μπορούσαν να είναι αντίθετες με, τις, ε, με τους κανόνες του ΠΟΕ και κατόπιν ε, πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν τη σημασία των μέλων με, των μέτρων όπως η κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων και τώρα μας είπατε ότι στόχος είναι να ζητήσετε από τα μέλη να ψηφίσουν με ειδική πλειοψηφία. Αν αποτύχει αυτό, ποια είναι η άλλη επιλογή. Ενισχυμένη συνεργασία τι να περιμένετε να αλλάξουν γνώμη. Ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Όπως ε, γνωρίζετε, κάναμε πολλό, πολλά σε νομοθετικό επίπεδο για να καταπολέμησουμε τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Χρησιμοποίησαμε τρόπο στα εργαλεία που είχαμε, κυρίως το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Υπήρξαν συζητήσεις με τις ΜΚΟ που έλεγαν ότι Έλεγα ότι, έλεγα ότι δεν υπάρχει φορολογικός παράδεισος στην Ευρώπη. Υπάρχει ανταλλαγή ε, ε, πληροφοριών και έχουν οι όλες οι χώρες υιοθετήσει το BEPS. Υπάρχει ένα σημαντικό διακύβημα που απομένει. Θέλουμε να υπάρξει ενθάρρυνση και διάλογος για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι υπηρεσίε μου έρχονται σε επαφή με τι εθνικέ διοικήσει και θέλουμε να στηρίξουμε τι εθνικέ αρχέ Το θέμα τη φορολογική επιθετικού του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ήταν στο επίκεντρο. Τι άλλαξε. Βλέποντας λοιπόν το φορολογικό σχεδιασμό στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, είναι ένας τρόπος να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη. Να δώσω ένα παράδειγμα και μόνο. Η Ολλανδία ήταν μία από τις χώρες με σύσταση που αφορούσε τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και, σχέσεις και χθε συναντηθήκαμε με Ολλανδού γερουσιαστέ που παρουσίασαν τι αλλαγέ που επέφερε η χώρα του, που ίσω δημοσιευτούν οι αλλαγέ ε, σήμερα, ήταν θεαματικέ. Ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τι ιδιαιτερότητε του φορολογικού του ε, συστήματο οι επιχειρήσει ε, για να έχουν πιο θετική φορολογική αντιμετώπιση. Αυτό δεν θα ίσχυε χωρίς την πίεση των ομοτήμων και χωρίς την κοινή μας ε, δράση και αυτό αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα. Η μεταρρυθμίση φορολογικής των ΗΠΑ εξακολουθούμε να το εξετάζουμε αυτό, έχουμε ανησυχίε για κάποια πράγματα. Η διά... Ε, λοιπόν, Υπάρχει ένα θέμα για τιμή κατάχρηση του φορολογικού νόμου και το θέμα ε, του IP για, το που, για την πνευματική ιδιοκτησία. Αυτά είναι κάτι που μας ανησυχεί, κυρίως για τις συνοριακές συναλλαγές, ε, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε αν συνάδουν τα μέτρα με τους κανόνες ΠΟΕ. Και ίσως να υπάρχει και εξα, εξαγωγική επιδότηση έμεση που απαγορεύεται από τον ΠΟΕ. Τα αντιμετωπίζουμε αυτά και στα πλαίσια διαλόγου με τους Αμερικανούς ομολόγους μας συναντήθηκα με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, τον Στίβεν Μανούτσι, στη Νέα Υόρκη τέλος Σεπτέμβριο. Εξακολουθούμε να συζητούμε και συνεχίζεται ο διάλογος. Τώρα, όσον αφορά το CCTB και άλλα ζητήματα, τι ελπίζω. Γνωρίζω ότι θα καταλήξουμε σε σε κάτι τελικό σε αυτή τη φάση. Έχουν απογοητευτεί εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που δεν ολοκληρώνουν τι συζητήσει, αλλά όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, υπήρξε μια πρόταση η οποία τελικά δεν πέρασε και είπα να αποσύρουμε, κάνουμε κάτι άλλο, να υποβάλουμε άλλη. Λοιπόν, πάντως προχωρούν τα πράγματα και ελπίζω ότι στο διάδοχό μου θα αφήσω μια κληρονομιά, αυτό το χαρτοφυλάκιο που θα μπορέσει να ολοκληρωθεί σε μερικούς μήνες. Αυτό ισχύει για το CCDB, για το ψηφιακό. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τη μάχη πάνω σε αυτά. Και για το ΦΠΑ κάναμε κάποια πρόοδο, αλλά δεν έγιναν όλα τα απαιτούμενα. Για να είναι ξεκάθαρος, η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία δεν πρέπει να μας καθυστερήσει, δεν θα πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία της πρότασης που ήδη έχει τεθεί επιτάπητος. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες το ταχύτερο δυνατόν πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεπε Κόφοντα, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε σήμερα εδώ να εκφράσω πρώτα απ' όλα την εκτίμησή μου για την καλή συνεργασία που έχουμε νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά τα επιτεύγματα αυτά και πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα πριν το τέλος της εντολής όπως ξέρετε κάτι το οποίο θα ήθελα να θέσω είναι ακριβώς αυτή η μειοδοσία όσον αφορά τον φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων αν δείτε τα τελευταία χρόνια έχει πέσει μέσω συντελεστής από το 25% στο 22% και η τάση είναι πτωτική. Οπότε τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να υπάρχει μια ελάχιστη αποτελεσματική φορολογία των επιχειρήσεων εντός της Ένωσης δεδομένου των περιορισμένων αρμοδιοτήτων όπως είπατε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις με το Συμβούλιο, διαβουλεύσεις με την ομάδα επαφής Πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη αναφέρατε τους φακέλους ε, και την ανάγκη πραγματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών. Τώρα λοιπόν με την ε, νέα οδηγία για την διοικητική συνεργασία θεωρείται ότι υπάρχουν οι απαραίτητες δομές ε, και δεν χρειάζεται συγκεντρωτισμός των δομών αυτών γιατί το σκάνδαλο αυτό όπως ακούσαμε συνεχίζεται υπάρχουν παρόμοια συστήματα σε κράτη-μέλη και σήμερα όπως ακούσαμε κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν για να σταματήσουν ναι ακούστε για το πρώτο θέμα η πρότασή μας για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων είναι η καλύτερη προσέγγιση και παρά το ότι το θέμα αυτό δεν αφορά συντελεστές αλλά έχει πρώτα απ' όλα στόχο να δημιουργήσει διαφάνεια και άρα δικαιότερο φορολογικό ανταγωνισμό. Βεβαίω, πέρα από αυτό υπάρχουν και κάποιοι κανόνες για να αποφεύγεται η κατάχρηση και οι επιχειρήσεις να μην μειώνουν υπερβολικά τους ε, φόρους τους. Ένας ελάχιστος συντελεστής όμως δεν είναι μέρος της ε, πρότασής μας, καθώς δεν έχουμε αρμοδιότητα, αλλά ελάχιστη πραγματική ε, φορολογία είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί με τα κράτη-μέλη. Ελάχιστη πραγματική φορολογία είναι η ιδέα ότι όλες οι εταιρείες θα πρέπει να πληρώνουν ένα ελάχιστο ποσοστό φόρου εντός ένωση, ανεξάρτητος του ύψους ε, που μπορεί να ποικίλει. Και έχει γίνει επίκαιρη τα τελευταία χρόνια δεδομένη τη ατζέντα τη Ευρωπαϊκής Ένωση για μια αποτελεσματική φορολογία και η Κομισιόν ήδη το 2011 είχε προτείνει μια ρήτρα ε, αποτελεσματική ε, φορολογία στο πλαίσιο τη οδηγία περί πνευματικών δικαιωμάτων αλλά τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταλήξει ακόμα τα συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ ε, της 15 ε, Δεκεμβρίου ζητούσαν ακριβώς ε, να υπάρξει μια συζήτηση του θύματος για ένα αποτελεσματικό επίπεδο φορολογίας των εταιρικών κερδών, όμως οι απόψεις ήταν αποκλίνουσες και όπως σας είπα η, έκθεση, η Κομισιόν με προετοιμάζει μια έκθεση που θα εξετάσει το θέμα και θα κάνει κάποιες συστάσεις για το σκανδαλοκόμ 6 και τα... Κοιτάξτε, κινήθηκα για να αλλάξουν οι το του παιχνιδιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την εποχή που ξεκίνησε το σκάνδαλο που ξέσπασε ε, έγιναν σημαντικές αλλαγές, ανταλλαγή αυτόματη των πληροφοριών, όχι κατόπιν αιτήματος, αυτό είναι ο κανόνας, και η διοικητική συνεργασία ενισχύθηκε και επεκτάθηκε. Συμπεριλαμβάνει ακριβώς και την αυτόματη ανταλλαγή υποχρεωτικά πληροφοριών για τους λογαριασμούς, για τις αποφάσεις επιφορολογικών των κατομελών, ε, tax ruling, ε, αναχώρα, παρόλο που θα θέλαμε να δημοσιευτούν ποιοι φόροι καταβάλλονται στι πολυεθνικέ και πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών και των αρχών κατά του ξεπλήματο χρήματο. Και αυτή η οδηγία ολοκληρώθηκε από, συμπληρώθηκε από νέε υποχρεώσει που προβλέπονται όσον αφορά τι δηλώσει για του ενδιαμέσου φορολογικού που δίνουν συμβουλέ που ίσω οδηγούν σε φοροδιαφυγή και φοροαπάτη. Δεν ξέρω τι θα ήταν αδύνατο να το σκάνδαλο σήμερα. Οι, οι πάντα έχουν μεγάλη φαντασία αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτού. Εν συνεχεία, μιλήσατε για μέτρα τα οποία είναι πολύ πρόσφατα. Δεν μπορώ να τα αξιολογήσω. Πιστεύω ότι ήδη σημειώνουν μια πρόοδο, σημαντική πρόοδο. Αυτή η πρόοδο δεν είναι το τέλο τη ιστορία. Θα πρέπει αναμφισβήτητα και από εσά ε, εξαρτάται η απόφαση να γίνουν συμπληρωματικέ προτάσει όσον αφορά βελτιώσει τη διοικητική συνεργασία, όσον αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την απάτη του ΦΠΑ και πιθανά αντίμετρα. Καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για να μειωθεί το περιθώριο απάτης ΦΠΑ, ειδικά μέσω των καρουσέλ. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις και θα ήθελα το σχολείο σας για την άποψή σας για τις δυνατότητες εφαρμογής αυτών των τεχνικών λύσεων και πώς έχουν τα πράγματα, πώς τα βλέπει η Κομισιόν. Οι τεχνικές ε, που έχω κατά το εξής είναι χωριστές ε, πληρωμές. Πληρωμή πηγαίνει εν μέρη στην τράπεζα και εν μέρη σε αυτόν ο οποίος λαμβάνει την πληρωμή. Δεύτερον, ηλεκτρονικό αρχείο όλων των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Και τρίτον, μια ιδέα που πρότεινε μια ομάδα ειδικών να χρησιμοποιήσουμε εικονικά νομίσματα για να πληρώνουμε τον ΦΠΑ. Κάτι το εξωτικό ομολογώ και θα ήθελα την άποψή σας. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά τον γενικό κανόνα μη κατάχρησης για τον υπολογισμό του εταιρικού φόρου που έχει περιληφθεί οπωσδήποτε στο πρώτο σχέδιο της έκθεσης και θα ήθελα να μου κάνετε μια πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής αυτού του κανόνα και ποια είναι τα αποτελέσματα. Για την απάτη του ΦΠΑ οπωσδήποτε ε, είναι καλοδεχούμενες τεχνικές προτάσεις που αναφέρατε αλλά η Κομισιόν θεωρεί ότι υπάρχει μια πιο συστημική ε, απάντηση για την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης και της απάτης καρουσέλ που είναι γύρω στο 50 δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα κάθε χρόνο για τα Υπουργεία Οικονομικών, δηλαδή να εγκριθούν οι προτάσεις που κάναμε για τις διασυνοριακές ε, συναλλαγές που κατά την άποψή μας πρέπει να θεωρούνται ε, εγχώριες. Και αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή και οπωσδήποτε βλέπουμε ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, πρόοδος. Η πεποίθησή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα οριστικό καθεστώς ΦΠΑ. Έχουμε πάρα πολύ καιρό ένα προσωρινό καθεστώς επί 25 χρόνια και πάμε για 26ο έτος. Οπότε ζητώ από τα κράτη-μέλη να σημειωθεί κάποια πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση ανεξαρτήτως ε, του χύψη πειράματος για την εστροφή της χρέωσης. Για το δεύτερο ερώτημα, καθώς ε, το ΑΤΑΤ 1 είναι μια πρόσφατη εφαρμογή, πρέπει να πω ότι δεν έχουμε ακόμα μία αξιολόγηση. Αλλά εάν οι υπηρεσίε μου έχουν κάτι πιο επικαιρό θα σας το στείλουμε. Σας ευχαριστώ. Το προσωρινό καθεστώς ΦΠΑ ε, κράτησε περισσότερο από την προσωρινή παραμονή των Σοβιετικών στρατημάτων στην χώρα μου. Λοιπόν, η έλισλαϊν για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε κύριε Μοσκοβισή για την εκ νέου εδώ παρουσία σας στην Επιτροπή μας. Αυτά τα χρόνια τα σκάνδαλα που ξέσπασαν έδειξαν σε αυτό τον τρελό φορολογικό ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ κρατών μελών. Είμαστε όλοι θύματα. Όλα τα κράτη-μέλη χάνουν, κερδίζουν μόνο αυτοί που καταφέρνουν να πληρώσουν σχεδόν μηδενικό φόρο. Εκφραστήκατε για δύο εργαλεία. Θα ήθελα μεγαλύτερη σαφήνεια όμω. Σε ποιο βαθμό βρισκόμαστε τώρα, σε ποιο σημείο είμαστε όσον αφορά το CCTV, ποια είναι τα εμπόδια για μια ταχεία έγκριση του σημαντικού αυτού μέτρου και όσον αφορά ε, το CBCR, άλλο σημαντικό εργαλείο, εξασφαλίσουμε ε, την καταστροφή των διαφόρων σχημάτων που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές για να, να αποφύγουν την ευρωπαϊκή φορολόγηση. Είναι σημαντικό αυτό. Ξεκίνησε ήδη τις εργασίες από αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανάλυση αντικτύπου ε, των κρατών μελών ε, και Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις αναπτυσσόμενες χώρες που βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από τη φοροαπηφυγή και τη φοροδιαφυγή των μεγάλων ομίλων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Ε, περιμένουν λοιπόν πάνω σε αυτό μια σαφή απόδειξη οι πολίτες ε, σε τι χρησιμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να ενοχλούν τα, κράτη, μελη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το τι γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μην ξέρουμε. Πιστεύω. Συμφωνώ μαζί σας ότι όλοι χάνουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει πολύ, υπάρχουν πολύ ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της, ε, των οικονομιών μας και οι φοροδιαφυγή και οι φοροαπάτες ε, μειώνουν την αξιοπιστία της Ένωσης, μειώνονται όμως και τα εισοδήματα και δημιουργείται δυσπιστία έναντι όλων των κρατών μελών αλλά και του συνόλου της Ένωσης. Λοιπόν, στον τομέα αυτό, όντω αποδεικνύει η Ευρώπη ότι λειτουργεί, γιατί έχουμε κάνει πολλά τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Κανείς δεν μπορούσε μεμονωμένα να επιλύσει τέτοιου τύπου προβλήματα. Αν όμως δεν μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, θα υπάρξει μεγάλη απογοήτευση από την κοινή γνώμη. Αυτό ισχύει για τα δύο θέματα που αναφέρατε. Για το CCCTB, η Ευρώπη πρέπει να έχει μια συλλογική προσέγγιση. Επιτέλους, να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο φορολόγησης των εταιριών. Αν θέλουμε μια πραγματική ενιαία αγορά. Έτσι οι επιχειρήσεις μας θα μπορούν να λειτουργούν ε, καλύτερα με μικρότερο κόστος και θα συμβάλλουμε παράλληλα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Συναντήθηκα με εκπροσώπους ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και συμφωνούν ιδιαίτερα με αυτό. Αλλά τώρα τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ξέρω ότι δεν θα καταλήξουμε το θέμα αυτό κατά την τρέχουσα θητεία, αλλά ελπίζω με τη στήριξη του Κοινοβουλίου να υπάρξει μια συμφωνία για κάποιες βασικές αρχές πριν το τέλος της θητείας, ούτως ώστε να αναλάβουν οι διάδοχοί μας και να ολοκληρώσουν ταχαίως. Να μην αποσυρθεί και πάλι το θέμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ξέρουμε ένα από τα θέματα που είναι πολύ δύσκολη συζήτηση είναι η ενοποιημένη φορολογική βάση. Γι' αυτό η Κομισιόν έκανε σε δύο φάσεις ε, την πρότασή της. Δεν ξεχνάω ότι το CCCTB έχει τρία C, όχι δύο. Για τις ε, αναχώρα εκθέσει τώρα. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο, αλλά και εμεί ω Επιτροπή, ενδιαφερόμεθα ιδιαίτερα. Η διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας. Γιατί ξέρετε ότι ορισμένες ε, πολυεθνικές ε, δεν είναι και τόσο ενθουσιώδος υπέρ της ε, διαφάνειας. Αλλά ορισμένες από την άλλη μεριά θεωρούν ότι πρέπει να ε, έχουν κάποια φορολογική στρατηγική. Και δεν κάνω δίκη προθέσεων για κανένα. Αλλά ορισμένοι θεωρούν ότι να αποκαλύψεις τις στρατηγικές σου προθέσεις αυτό σε αποδυναμώνει. Η διαφάνεια όμω ισχύει για όλου. Ισχύει για τι κυβερνήσει, ισχύει για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, άρα ισχύει και για τι επιχειρήσει και τι πιέζει. Δεν μπορούμε να αντιπαραθέτουμε την διαφάνεια στην ανταγωνιστικότητα. Μετά από μελέτη αντικτύπου, μετά από εσωτερική συζήτηση, μετά από δημόσια διαβούλευση, η Κομισιόν και επίση φυσικά προ την την κατεύθυνση, διατύπωσε μια πρόταση που είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, αλλά θα ήθελα να πάμε πιο γρήγορα να ολοκληρώσουμε αυτό που αναλάβαμε. Νομίζω ότι θα είναι και δική σας ε, παρακαταθήκη στο επόμενο κοινοβούλιο να προχωρήσει πιο γρήγορα. Εάν δεν προχωρήσει στο Συμβούλιο, να είστε σίγουροι ότι δεν φταίει γι' αυτό αδράνεια από πλευράς μας. Ο Βολφ Κλίντ. Κύριε Επίτροπε, καταπολεμάτε τις φορολογικέ απάτε και την φορολογική εγκληματικότητα. Θαυμάσιο και σας συγχαίρω. Αλλά η δίκαια φορολόγηση τώρα. Θέλετε να φορολογηθεί ε, η ψηφιακή δραστηριότητα. Αυτό νομίζω είναι λάθος, γιατί έχετε λάθος στοιχεία. Βασίζεστε σε μια εξομοίωση που έκανε το Ινστιτούτο ZTV του Πανεπιστημίου του Μάνχαϊμ. Πού κατέληξε στο συμπέρασμα αυτή η μελέτη λοιπόν, ότι οι ψηφιακές ε, επιχειρήσεις πληρώνουν 9,5% ενώ οι παραδοσιακές ε, μόνο περίπου 30% φόρου. Αλλά ήταν μια εξομοίωση. Και ο επικεφαλής ε, της μελέτης αυτής έχει απομακρυνθεί από τα αποτελέσματα εντωμεταξύ. Δεν θέλει να αναφέρει το όνομά του σε σχέση με τη μελέτη αυτή και έκανε και δημοσιεύσεις που την καταρρύπτουν. Και λέει καθαρά ότι η Κομισιόν δημοσιεύει ψευδή δεδομένα. Λέει ότι η πραγματικότητα είναι ότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις φορολογούνται 20% και οι μη ψηφιακές 28 με 29%. Εάν λοιπόν ε, υιοθετήσετε αυτήν την φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών σε αυτή τη βάση, θα κάνετε μεγάλο λάθος. Γιατί θα αλλάξετε την αρχή την οποία ε, εφαρμόζουμε για δεκαετίε ότι τα προϊόντα φορολογούνται, τα, μάλλον τα κέρδη συγγνώμη, φορολογούνται εκεί που, προκύπτει, που παράγεται το προϊόν και η φορολόγηση των πωλήσεων γίνεται εκεί που γίνονται οι πωλήσει. Οι αμερικανικέ επιχειρήσει θα θεωρήσουν ότι είναι στην πράξη δασμό αυτό και δεν θα το δεχθούν ε, εύκολα. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν αντίμετρα από πλευρά του. Άρα θα έχουμε δυσχέρειε αργά ή γρήγορα μεταξύ Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών. Μα γιατί ακολουθείτε αυτήν την ε, οδό, χωρίς να είστε σίγουρος ότι είναι σωστά τα στοιχεία. Δεν είναι μόνο αυτή η μελέτη που τώρα αφισβητεί τον εαυτό και το Ινστιτούτο Οικονομικών Μελετών της ε, Κομεχάγης, ένα Ινστιτούτο στην, ε, και στο Μόναχο και άλλα επιστημονικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα λένε ότι η βάση υπολογισμών σας είναι λανθασμένη. Άρα κάνω έκκληση Προσέξτε, μην ορμήσετε σε λάθος κατεύθυνση. Κοιτάξτε, τα στοιχεία μπορούν να αμφισβητηθούν οπωσδήποτε με τον ένα ή με κάποιον άλλον τρόπο. Η συναδελφός μου, η Μάργαρετ Βεστάγκερ, έκανε κάποιες έρευνες και κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα ότι η χύψη η εταιρεία, δεν θα την πω τώρα, την ξέρουν όλοι, όχι επειδή το πραγματικό ποσοστό ήταν 9% αλλά 0, κάτι ο πραγματικός συντελεστής. Ε, πολύ μεγάλε εταιρείε λοιπόν πληρώνουν ε, ελάχιστο ή καθόλου φόρο εκεί που δημιουργούν αξία και κέρδη. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτή η φορολογία είναι θεμητή. Μετά βεβαίω επαφίεται στα κράτη-μέλη να το συζητήσουν όπως είπα. Όπως είπα αυτή στιγμή σήμερα μια εβδομάδα πριν το ΕΚΟΦΗΝ δεν βλέπω κάποια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει βεβαίως και η πρόθεση να φορολογούμε τα κέρδη, όχι τα έσοδα, αλλά πρέπει να στείλουμε και ένα σύμβολο της πολιτικής μας βούλησης, γιατί προφανώς ε, είναι κάτι το αναμενόμενο. Θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και τι συμπεράσματα θα πρέπει να βγάλουμε. Αλλά κάτι στο οποίο νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ένας κίνδυνος. Εάν δεν έχουμε κοινό, κοινή προσέγγιση θα υπάρχουν ε, εθνικές προσεγγίσεις και αυτό είναι το χειρότερο για την εσωτερική αγορά και τις εταιρείε μας. Για το όλο το οποίο αναφέρατε τις είπα και αυτό συζητάμε με τον κύριο Μινούτσιν και ε, με τον κύριο Ρώσο το συζήτησα στην Ουάσιγκτον πριν από έξι μήνες στις προηγούμενες συνεδριάσεις του ΔΕΛΤΕΝΤΑΦ. Κοιτάξτε, ο Υπουργό των Οικονομικών τον ΗΠΑ συμφωνεί μαζί μας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει ακριβώς να το αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο του ΩΣΑ. Το ερώτημα είναι ακριβώς εάν η ΕΠΑ θα επιδείξει μια ηγεσία ή όχι. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν δύο προτάσεις και όχι μία. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ασκήσει κάποια ηγεσία μετά. Με τον Γουλμπορός ήταν κάπως πιο δύσκολα τα πράγματα. Και έχω να πω δύο πράγματα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι το θέμα είναι να φορολογήσουμε Google, Amazon, Facebook και Apple. Δεν αφορά τέσσερις εταιρείε το θέμα, αφορά εταιρείε οι οποίες έχουν ε, έσοδα άνω των 750 δισεκατομμυρίων παγκοσμίω, 50 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι φόρος για αυτές τις εταιρείε, ούτε στρέφεται κατά τον ΙΠΑ. Βεβαίως βλέπουμε ότι προφανώς υπάρχουν ε, ίσως 150 εταιρείες ε, που μπορεί να τι αφορά το θέμα. Από αυτές οι μισές ε, πιθανώς θα είναι αμερικανικές γιατί έχουν ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Οι υπόλοιπε όμως είναι ευρωπαϊκές και από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι λοιπόν προστατευτισμός, δεν στρέφεται κατά τεσσάρων εταιρεών, ούτε κατά τον ΙΠΑ. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει και κάποιο αντικείμενο για αντίπεινα. Και θα τα συζητήσουμε αυτά με τους Αμερικανούς φίλους μας και στους G20. Όταν θα μιλήσω με το Υπουργείο Οικονομικών στους G20 και, και νομίζω ότι έχουμε γενικά μια αρμονική συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Σβέν Γκίγκολτ για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς εσάς κύριε Επίτροπε για τα επιτεύγματά σας. Μπορούμε να πούμε ειλικρινά ότι σε κανέναν άλλο τομέα νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως επετεύχθη τόσο μεγάλη πρόοδο στην τελευταία πενταετία σε κανένα άλλο τομέα από ότι στον τομέα τη φορολόγηση και το ξέπλυμα χρήματο. Το ξέπλυμα χρήματο δεν είναι αποκλειστικά δική σα ευθύνη. Συνεργάζεστε με την Επίτροπο την κυρία Θα πρέπει να δείτε ότι ε, δεν είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες. Δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένοι. Χθε συγκλονιστήκαμε με αυτά που ακούσαμε στην ακρόαση. Όλοι οι παρόντες συμφώνησαν από αυτού, ανεξάρτητα από την πολιτική επιλογή. Η ακρόαση COMEX και οι δημοσιογράφοι απεκάλυψαν ότι παρά τις κοινέ μας ε, προσπάθειες, η COMEX και η COMCOM ε, συνεχίζεται. Είπαν σαφώς ότι πρόκειται περί ευρωπαϊκού σκανδάλου. Υπάρχει μεγάλη διασυνοριακή δραστηριότητα και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να κινηθούμε προς ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομία και ευρωπαϊκές ε, φορολογικές δυνατότητες σε διοικητικό επίπεδο. Δεν το έχουμε ακόμα αυτό. Είναι συγκλονιστικό, Επίτροπε, διότι περισσότεροι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών δεν το σχολίασαν καν αυτό. Εσείς ε, με προσοχή κάνατε κάποια σχόλια και κατά το παρελθόν μιλήσατε πολύ προσεκτικά για το θέμα. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα κινηθείτε όσον αφορά το cum και το cum ε, θα μπορούσατε να δρομολογήσετε έρευνα από τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Αρχές δυνάμει του άρθρου 22.4 των κανονισμών περί των Ευρωπαϊκών ε, Δημοσιονομικών Αρχών ε, Οικονομικών Αρχών. Μπορείτε να ερευνήσετε αυτό το σκάνδαλο όπως ερευνήσατε κι άλλα και να κάνετε τις σχετικές προτάσεις. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε να αναλάβει τα καθήκοντά της η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει οι πολίτες ε, πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές να δούνε μια στεναρή και ξεκάθαρη απάντηση. Και βασίζομαι σας. Ευχαριστώ κύριε Γκίγκολντ. Είμαι πολύ ευαίσθητος όσον αφορά αυτό το... τις ευχαριστίες σας. Θυμάμαι τόσο στο τέλος θητείας την αρχή και τη συζήτηση που είχαμε όπου ετέθη το θέμα της επικύρωσης εκλογής μου στη θέση του Επιτρόπου. Λοιπόν, έκτοτε συνεργαστήκαμε πολύ καλά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Ήταν ομαδική συνεργασία η εργασία που κάναμε για το σκάνδαλο. Έδρασα για να αλλάξουν οι κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μεταξύ άλλων θα παρατήσετε τη η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία επεκτάθηκε και ενισχύθηκε σημαντικά διότι προβλέπεται αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών πλέον όσον αφορά τους, τους λογαριασμούς οικονομικούς και έχουμε και νέες διατάξεις όσον αφορά τις για τους ε, φορολογικούς ενδιαμέσους που δίνουν συμβουλές που μπορεί να οδηγήσουν φοροδιαφυγή ή σαπάτη. Για την παρακολούθηση τώρα, την εποπτεία των συναλλαγών και θα πρέπει να επιβάλλουν τους φόρους στα κράτη-μέλη μέσω της φορολογικής τους νομοθεσίας και παρακολουθεί από κοντά τους σχετικούς ε, βάσει των κανόνων περί συνεργασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται στην ανταλλαγή πληροφοριών για τα φορολογικά μεταξύ των κρατών μελών πέρα από αυτού, από την αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών που επεκτάθηκε σημαντικά, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν επίση αυθόρμητα πληροφορίε που όταν θεωρούν ότι υπάρχει απώλεια φόρων σε άλλα κράτη-μέλη, και ενθαρρύνω να το κάνουν αυτό τα κράτη-μέλη και να κινούνται πάρα πολύ γρήγορα για να αποφευθούν απάτε. Τακτικά δίνουν στατιστικά στοιχεία στι υπηρεσίε μου και οι υπηρεσίε αξιολογούν κατά πόσο εφαρμόζονται οι κανόνε περιδικητική συνεργασία. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η ανάλυση το πρώτο τρίμηνο του 2019, πριν από τι ευρωεκλογέ, ε, θα μπορούσε να έχουμε μια πρόταση για μελλοντικέ βελτιώσει, εάν θεωρηθεί κάτι τέτοιο αναγκαίο. Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω στη θέση των ε, αρμοδίων αρχών για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα. Όσον αφορά το φορολογικό τομέα, στα σκάνδαλα ε, έχουμε, έχουμε μακροσκελή κατάλογο φορολογικών ε, απατών. Υπάρχει λοιπόν ε, λόγω της εξυπνάδας, της ανευθυνότητας ε, κάποιων της εξυπνάδας αυτών που θέλουν να εξαπατήσουν μη εφαρμογή σωστά του νόμου και ενώ που υπάρχουν νομοθεσία, ελλείψεις στον φορολογική συνεργασία για τα θέματα τα φορολογικά ε, πριν τα μεταρρυθμίσουμε, υπήρξαν, υπήρξε μια κροσκελή κατάλογο σκανδάνων φορολογικών. Και αξιολογούμε λοιπόν το πλαίσιο τη διοικητική συνεργασία που υπάρχει βάσει των νέων κανόνων που σταδιακά υλοποιούνται. Αυτό το σκάνδαλο ακόμα και είναι. Ε, ε πρέπει να οδηγήσει την αξιολόγηση των προβληματισμών. Να πω πρώτα απ' όλα ότι θα λάβουμε υπόψη παρακολουθώντας του Ξύνεγγι, τα συμπεράσματα και τη δική σα έρευνα. Ε, δεύτερον, ε, λαμβάνοντα υπόψη το εύρο του σκανδάλου, χρειάζεται ενδελεχή έρευνα Ίσως να είναι κάτι αναγκαίο και έτσι θα κάνουμε τις δικές μας έρευνες και θα προχωρήσουμε περαιτέρω τις δικές μας εργασίες αν αυτό καταστεί αναγκαίο από την ενδελεχή έρευνα. Για το EFTD, Πιέρ Νίκολα Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ. Επίτροπε, θα ήθελα να στραφώ στους φορολογικούς παραδείσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σπίτι μας η φορολογική παράδειση που είναι αυτή, το είπατε πριν αλλά το υπενθυμίσατε και στην οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση της Ένωσης τον περασμένο Μάρτιο και το Βέλιο, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και κάτω χώρες είπατε ότι χρησιμοποιούνται φορολογικό σχεδιασμό επιθετικό όπως αποκαλείται και χάρη σε αυτή την επιθετικότητα αυτές οι χώρες είναι πιο πονηρές, πονηρές χώρες και καταστρέφουν την εσωτερική μας αγορά διότι από τη μία πλευρά προσελκύουν εταιρείε άλλων χωρών που θέλουν να ξεφύγουν από τα κεφάλαιά τους και γίνεται και αθέμητος ανταγωνισμός ε, έναντι των εταιριών που πληρώνουν υψηλότερους φόρους εντός των χωρών ε, που εδρεύουν. Είπατε ότι δεν προτίθεστε να δακτυλοδείξετε αυτές τις χώρες, αλλά φαίνεται όμως να ζουν σε μια αντίστροφη πραγματικότητα. Από τη μια πλευρά αυτές οι χώρες ε, βραβεύονται ουσιαστικά, διότι δεν επιβάλλονται κυρώσεις, ενώ ε, έμεσα κάνουν να πληρώσουν οι άλλες χώρες που σέβονται αυστηρά τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Φαίνεται ότι λόγω της ομοφωνίας όλα είναι αδύνατα να βρεθούν λύση. Τώρα στο τέλος της θητείας αυτός ο κανόνας περί είναι κάτι που αμφισβητείται. Καλή αργά παρά ποτέ ερώτηση που κάνω εγώ, που κάνουν πολλοί πολίτε και εγώ. Τι κάνετε συγκεκριμένα, όχι τι θα γίνει, τι κάνετε. Δεν μιλώ για καλέ προθέσει. Τι κάνετε συγκεκριμένα για να εξαλειφθεί η μεγάλη αδικία, να επιβληθεί μια ισότιμη, χωρί εξαιρέσει φορολόγηση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Σε ποιο σημείο είναι η, ε, η όλη ε, εφαρμογή αυτών των σχετικών διατάξεων να αποφευθεί αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι επίμαχο το θέμα δεν θα σας διαφεύγει, δεν διαφεύγει ότι άλλες αρχές, ΜΚΟ, είχαν επεξεργαστεί καταλόγους φορολογικούς παραδείσους που καμιά φορά εμφανίζονται και ευρωπαϊκές σημαντικές χώρες και υπάρχουν και μελέτες πανεπιστημιακές που προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Θεωρώ ότι όταν βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό πλαίσιο, είναι ένα πλαίσιο πολιτικό και όταν δρομολογούμε δράσεις, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από ακριβείς ορισμούς. Τι είναι ένας φορολογικός παράδεισος. Σχετικά με αυτό έχουμε καθορίσει τις δικές μας προσεγγίσεις όταν επεξεργαστήκαμε μαζί με το δοτικό κώδικα έναν μαύρο κατάλογο, μια μαύρη λίστα που καταρτήσαμε για φορολογικών παραδείσων όσον αφορά τις εταιρείε. Λοιπόν, λοιπόν, και πού οδηγηθήκαμε από αυτό. Θέλαμε να δούμε αν οι χώρες υιοθετούν ή όχι τους κανόνες BEPS και το δεύτερον εάν μεταξύ τους ανταλλάσσουν πληροφορίες ή όχι. Και τι διαπιστώσαμε. Εάν παρακολουθήσουμε αυτόν τον ορισμό, που δεν αφορά όλο τον πλανήτη, διότι βρίσκεται περίπου, βρίσκονται 75 χώρες στο, στο γκρίζο, στην γκρίζα λίστα και 5 στη μαύρη λίστα που δεν αμεληταίο, δεν υπήρχαν χώρες τη Ευρωπαϊκή Ενώση που θεωρούνται φορολογική παράδειση και γι' αυτό στην αρχή όταν κάναμε το screening, τη διήθηση, τη λεπτομερή των χωρών για να δούμε ποιες χώρε ε, θα μπορούσαν να μπουν στον κατάλογο. Δεν είχαμε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη μαύρη λίστα. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ορισμό, δεν υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω έχω επίγνωση ότι υπάρχουν κάποιε πρακτικέ που αυτέ οι πρακτικέ δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτέ. Ε, το αλλάξαμε, αλλάξαμε την προσέγγιση, εκμεταλλευτήκαμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο ούτω ώστε να ασκήσουμε φιλική πίεση μέσω διαλόγου, αλλά στεναρή πίεση παρόλα αυτά, έναντι κάποιων χωρών και λέμε ότι ακολουθούν πρακτικές φορολογικό επιθετικό σχεδιασμό ή πρακτικές που ενθαρρύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και αυτές οι χώρες κατονομάστηκαν. Εγώ δεν πέρασα το καλύτερο κοφή μου εκείνη την ημέρα, δεν ήταν και πιο καλή και ευχάριστη συνάντηση αυτή. Απάντησα στενερά και με ηρεμία στις ερωτήσεις και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και σημείωσα όσον αφορά τις κατοχώρες το θέμα. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα. Δεν ήταν άχρηστη πίεση διότι οδηγούσε σε αλλαγή των συμπεριφορών και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο, αυτό το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε με στεναρό και φύη τρόπο και στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εξαμήνου για πρώτη φορά κατόπιν παρότησής μας ε, εισήχθη η φορολογική πτυχή και οι υπηρεσίες μας βλέπουν, ε, συναντούν τις φορολογικές αρχές και τους συμμετέχοντες και μπαίνει αυτή η διάσταση και ο στόχος είναι να έχουμε μια κοινή ανάλυση του διακυβεύματος. Από τη στιγμή που έχουμε κοινά συμπεράσματα και ανάλυση να αλλάξουμε τις πρακτικές που ακολουθούνται. Μάριο Μποργέτσιο για το ENF. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στις απαντήσεις σας είδα ότι υπάρχει μεγάλη προσοχή και σύνεση όσον αφορά να εντοπιστούν οι αρνητικοί ε, ε, πρωταγωνιστές του ΚΟΜΕΞ. Ήσασταν πολύ γενικόλογος. Αλλά κατά την άποψή μου παραλείψατε σκόπιμα Εμεί βέβαια οι πολιτέ χαλιών είμαστε πολύ καχύποπτοι. Ότι, να πείτε ότι οι μεγάλες τράπεζες είναι οι πρωταγωνιστές ε, από ό,τι λένε οι έρευνες, τα αποτελέσματα των ερευνών του γερμανικού δικαστικού κλάδου και από την έρευνα που έκαναν οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι, οι ερευνητές δημοσιογράφοι, διαπίστωσαν αυτό. Και στην αίθουσα είπαν ότι το σκάνδαλο δεν ε, αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά. Αντίθετα, λαμβάνοντας υπόψη και την τεράστια κλίμακα του σκανδάλου και τη ζημιά που υπέστησαν κάποιες χώρες. Που είναι σημαντική ζημιά και ε, για μια χώρα όπως η Ιταλία, 4,5 δις ευρώ. Και είπαν οι εμπειρογνώμονες ότι σε χώρες όπως η Ιταλία το σκάνδαλο συνεχίζεται. Συνεχίζεται η ζημιά δηλαδή. Ερώτηση. μήπω θεωρείτε ότι ήταν αδύναμη η αντίδραση. Ήσασταν ήδη υπουργό οικονομικών όταν ε, ε, εφαρμοζόταν το σκάνδαλο. Και τώρα αυτούς τους μήνες σαν ε, Ευρωπαίος Επίτροπος δεν θα πρέπει να μιλήσετε με σαφή φωνή. Μόνο όταν θέλετε να μαστιγώσετε την Ιταλία μιλάτε με δυνατή φωνή που παραβίασε έναν κανόνα που παραβιάστηκε στην περίπτωση της Ισπανίας, της Γαλλίας Μήπως εκεί ήσασταν πολύ μεγαλόφωνος. Μήπως εδώ πέρα ε, δεν, αποφεύγετε να κατονομάσετε αυτούς που πρωταγωνιστούν σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Μπορεί να το εξηγήσετε αυτό. Εσείς σαν Ευρωπαίος Επίτροπος πρέπει να υπερασπίζεστε και τους αποταμιευτές ε, των κρατών μελών, ξεκινώντας από τη χώρα μου, που δεν πρέπει να ποινικοποιείται που αποφάσισε να αλλάξει πολιτική και να μην υπακούει σε κανόνες που όπως έλεγε ο Τζοβάνι Τζολίτη, μεγάλος πολιτικός της χώρας μου, που δεν ανήκει στη δική μου προσέγγιση, αλλά ήταν μεγάλος πολιτικός, έλεγε ότι οι κανόνες για τους άλλους εφαρμόζονται και για τους φίλους ερμηνεύονται. Εγώ έχω την εντύπωση ότι όσον αφορά τα θέματα, τους κανόνες, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ερμηνεύει κατά το δοκούν όπως βολεύει. Αναφερθήκατε σε άλλα θέματα, όχι μόνο σε φορολογικά θέματα. Με επιτρέπετε να κάνω έτσι μια διευκρίνηση που δεν θα ε, ότι δεν θα ήθελα ποτέ να θεωρήσω τους φίλους μου τους, και δεν θα περιέγραφα ποτέ τους φίλους μου τους Ιταλούς ως ε, εμπόρους ε, χαλιών ανθρώπους που, παρα, που παζαρεύουν δηλαδή ε, ήθελα να πω κάτι άλλο ότι δεν ε, μην ανησυχείτε, το θεωρώ αυτό σαν κομπλιμέντο, διότι είναι πάρα πολύ καλή έμπειρη. Και εγώ είμαι από οικογένεια, κατάγομαι από οικογένεια εμπόρων. Euh, Και εγώ είμαι από οικογένεια εμπόρων. Αλλά δεν πουλάγανε χαλιά, πουλάγανε πουλόβερ. Πλεκτά. Μου αρέσει πολύ το εμπόριο. Αλλά κοιτάξτε, αυτό που είπα προηγουμένω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ε, εκπτώσει ε, με του κανόνε. Κάνει εκπτώσει στι τιμέ, αλλά όχι στου κανόνε. για το Σταύλο Κουμέξ. Δεν θα εκφραστώ ε, ε, σοφρόνος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζω, όπως είπε και ο Σβέν Κίκολ, δεν έχει όλες τις πληροφορίες και ούτε δυνατότητα να τις έχει αυτή τη στιγμή σήμερα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμεθα με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις με βάση την, ε, τα στοιχεία που έχουμε από τα μέσα και τονίζω ότι αν πρέπει να προσαρμόσουμε την διοικητική συνεργασία ή να ξεκινήσουμε ε, έρευνε, θα το κάνουμε. Είπατε ότι ήμουν υπουργό Οικονομικών στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι η χώρα της οποίας ήμουν υπουργό Οικονομικών ήταν ε, η χώρα που ήταν κυρίω ή περισσότερο ένοχη στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών με βάση ε, τα μέσα μάλλον μια άλλη μεγάλη χώρα έκανε τέτοια πράγματα, αλλά κοιτάξτε, κάντε εσεί τη δουλειά σας και θα κάνουμε και εμείς τη δική μας. Νομίζω ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων μας θα μας επιτρέψει να είμαστε αποτελεσματικοί. Και φυσικά σας ακούμε και έτοιμοι να αντιδράσουμε σε αυτό που μας λέτε. Και κατάλληλα κύριε ε, συνάδελφε. Δεν δράει η Επιτροπή ποτέ με παροπίδες. Όχι, είμαστε πάντα επικοδομητικοί. Κοιτάξτε, όπω είπατε και στην αρχή, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Δεν είναι η Επιτροπή κατά τη Ρώμη. Η Επιτροπή δεν είναι μόνη τη. Η ε, Επιτροπή δρά με βάση του κανόνε σε ένα οικοσύστημα. Και εγώ ήμουν πάντα στα πλαίσια τη Επιτροπή, πάντα υπέρ τη ε, ευελιξία. Αλλά υπάρχουν και 18 για την Ευρωζώνη, Υπουργοί Οικονομικών, που και εκείνοι έκαναν πολλέ προσπάθειε κατά τη διάρκεια τη ε, κρίση για να εφαρμοστεί το σύμφωνο και το σύμφωνο για αυτού είναι ο κανόνα και πρέπει να εφαρμοστεί. Εγώ είμαι απόλυτα ευέλικτο. Ε, είμαι πάντα υπέρ του διαλόγου. Ε, δεν είναι τυπικό πράγμα ο διάλογο, ουσιαστικό, αλλά εντό των κανόνων. Μπορούμε να, τις, ε, να τους εφαρμόσουμε με το πιο έξυπνο, το πιο λεπτό τρόπο κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους κανόνες. Εγώ ε, ως Επίτροπος της Ένωσης δεν ε, είναι ο ρόλο μου να ε, αγνοώ, αλλά να εφαρμόζω του κανόνε, αλλά προ το κοινό συμφέρον, ε, επιδιώκοντα την εξέβρεση λύσεων. Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για την μόνιμη καλή σας διάθεση να έρχεστε εδώ. Θα ασχοληθώ με διεθνή συνεργασία. Ο Άγχελ Γκουρία ε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ ήταν μαζί μου σε μία εκδήλωση την προηγούμενη Παρασκευή. Αναφερθήκατε στο G20. Ξέρετε ότι θα γίνει μια συνεδρίαση στο Buenos Aires ε, αυτή τη βδομάδα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς εργάζεστε στα πλαίσια της ομάδας για την ε, διεθνή συνεργασία. Βλέπω ότι είστε πολύ ενομερημένοι για τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Πριν από την ακρόασή σας είχαμε μία έκθεση όπου προτάθηκε να υπάρξει μια υποεπιτροπή της ΕΚΟΝ για να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Η ερώτησή μου ασχολείται με κάτι που αναφέρει αυτή λοιπόν η έκθεση που συζητήσαμε προηγουμένως. Συζητάτε τις διμερείς ε, φορολογικές συμφωνίες που κάνουν κάποιες χώρες με τρίτες χώρες με στόχο να εναρμονιστεί το φορολογικό πλαίσιο. Και επίση αναφερθήκατε στο εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ επιτυχημένη δυναμική ε, εμπορικών συμφωνιών. Ολοκληρώσαμε τον Καναδά, την Ιαπωνία, το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, το Μεξικό. Ε, διαπραγματευόμεθα με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Τι σημασία αποδίδεται στα πλαίσια αυτών των εμπορικών συμφωνιών και συμφωνιών συνεργασία στην σωστή φορολογική διακυβέρνηση και ε, ρήτρε για την αμοιβαία εφαρμογή τέτοιων διατάξεων. Ευχαριστώ πολύ. Και ρητρών. Ευχαριστώ πολύ. Είστε πάντα ακριβείς, αλλά και κάνετε ερωτήσει που πάνε μακριά, αγαπητέ συνάδελφοι. Συνεργαζόμαστε με τον ΩΣΑ υπό την αιγίδα του G20. Και από την αρχή έχω τονίσει ότι οι Ευρωπαίοι από την αρχή ασχολήθηκαν με τα BEPS. Θυμάμαι ότι ο Ισπανό Υπουργό Οικονομικών, ο Δεγίνητος, ήταν εκεί από την πρώτη συνάντηση στο πλάι του Γενικού Γραμματέα του ΟΣΑ με τον οποίο έχουμε, με τον οργανισμό του, έχουμε μόνιμες σχέσεις. Είτε για τα ίδια το BEPS, την καταπολέμηση της φοραπάτης, αλλά και τη φορολόγηση της ψηφιακής δραστηριότητας ή για τη διαδικασία ε, κατάρτισης καταλόγων φορολογικών παραδείσων συνεργαζόμεθα πλήρω με τον ΟΣΑ, αλλά θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα. Γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα ότι είμαστε μια πολιτική ένωση και μια εσωτερική αγορά. Έχουμε λοιπόν μια παρουσία στην παγκόσμια σκηνή. Για τις δύο οδηγίες ε, για την ε, φοροαποφυγή, εμείς πήγαμε παραπέρα. Πήγαμε ε, σε κάτι που θα αποκαλούσα BEPS συν ή ο συν. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Ήμασταν οι πρώτοι που εγκρίναμε τις δράσεις του ΩΣΑ, οι πρώτοι που τις ε, μεταφέραμε στην οδηγία κατά της φοροδιαφυγής και οι εργασίες για την φορολόγηση της ψηφιακής ε, δραστηριότητας θέλουμε να είναι κάτι στο οποίο είμαστε πρωτοπόροι. τι συστάσει μπορούμε να κάνουμε για τις διμερείς ε, συμφωνίες. Ναι, όπου είναι αναγκαίο το κάνουμε. Για παράδειγμα, η ψηφιακή παρουσία. Επιμένουμε πολύ σε αυτό. Ξέρετε, ότι μας ενδιαφέρει πολύ. Για το διεθνές εμπόριο τονίσατε ότι η Επιτροπή σα, ε, συγγνώμη, η δική μας Επιτροπή ενδιαφέρεται για το ελεύθερο εμπόριο. Θα πάει και ο πρόεδρος Γιούγκερ στο μαζί μου, θα πάω μαζί του μάλλον στο Buenos Aires, για να στείλουμε το μήνυμα ότι ο προστατευτισμός δεν είναι λύση. Η πολυμερής ε, προσέγγιση είναι η καλύτερη. Θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε τον ε, ΠΟΕ, όχι να τον καταστρέψουμε και βεβαίω οι κανόνε ε, καλή φορολογική διακυβέρνηση είναι αποτελεσματικοί και η αμοιβαιότητα είναι πολύ σημαντική. Την αναμένουμε από όλου του εταίρου μα. Είναι μια βασική αρχή που αναφέρεται σε όλα τα σχέδια συμφωνιών που συζητάμε με του εταίρου μα. Δεν ξέρω αν το λάβατε υπόψη. Στην ε, μελλοντική συμφωνία με το Ηνωμένο Εμπόριο, που δεν είναι ακόμη συμφωνία ελευθερών εμπορίου, εάν ε, βεβαίως εγκρίνουν τον Brexit, θα εφαρμόσουν τους κανόνες σωστή φορολογική διακυβέρνησης. Δεν θέλουμε στα σύνορά μα να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει ένα κράτος που ε, δεν θα τηρεί αυτούς τους κανόνες. Ε, το επιδιώκει και το Ρωμένο Βασίλειο που πάντα ήταν στο πλευρό μας ως πολύ ενεργός εταίρος σε όλες τις ζητήσεις για τον ΠΕΠΣ e και τους φορολογικούς παραδείσους. Τελευταίος ομιλητής ο Πολ Τάνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Κοιτώντας την περίοδο που πέρασε είδαμε πολλές αλλαγές και νομίζω πως είχατε και εσείς μια μεγάλη συνεισφορά σε αυτές. Περισσότερα άλλαξαν τα τελευταία πέντε χρόνια από ότι τα προηγούμενα 50. Είδαμε κάποια ευρωπαϊκή συνεργασία στην φορολογία, η οποία βεβαίως χρειαζόταν πολλές ε, πρωτοβουλίες έχουν ε, ξεκινήσει, όχι από εσάς, δεν έχουν αποδώσει όλες, αλλά τουλάχιστον κάτι ξεκίνησε. Κάτι είναι και αυτό. Αυτό το οποίο είπε ο Βολφ Κλίντς ε, επίσης. Εγώ θα το έλεγα διαφορετικά. Αυτό το οποίο μας λείπει εδώ πέρα και στην Κομισιόν είναι τα δεδομένα και η δυνατότητα ανάλυσης. Συζητάμε τώρα ακριβώς ε, το DST και τις διάφορες ε, των φόροψιακών υπηρεσιών και τις διάφορες ε, παραλλαγές του. Θα θέλατε να δείτε και τις υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο συλλογής δεδομένων και ανάλυσης ε, που θα μας βοηθούσαν στην χάραξη φορολογικής πολιτικής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο νομίζω θα μας ε, βοηθούσε. Γιατί έχουμε ένα δημοσιονομικό συμβούλιο και όχι ένα φορολογικό συμβούλιο, παραδείγματο χάρη. Αυτό θα ήθελα να σκεφτείτε. Το δεύτερο, επίσης, αναφέρθηκε η ιδέα της μαύρης λίστας για τα μη συνεργαζόμενα κράτη είναι κάτι το πολύ ισχυρό αλλά σε τελική ανάλυση ε, έχουμε μόνο πέντε χώρες τι, τι σημαίνει αυτό και λέμε τώρα ότι αποκλείουμε τους φορολογικούς παραδείσους εντός της Ένωσης και προσπαθήσατε να το αντιμετωπίσετε. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό, γιατί τα κράτη-μέλη και αυτά έχουν κάποια αρνητική επίδραση. Σας ευχαριστώ κύριε Τάγκ και ήθελα να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για την τεράστια δουλειά που κάνετε για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων και ελπίζω και η δική σας εκληρονομιά να είναι ότι ακόμα και αν δεν ολοκληρωθεί ο φάκελος θα είναι έτοιμος και ελπίζω να συνεχίσετε να παλεύετε για το θέμα αυτό και την μέρα που θα περάσει αυτό. Νομίζω πρέπει να τιμήσουμε και εσάς. Μετά για τα ερωτήματα που αναφέρατε για τα δεδομένα, συμφωνώ μαζί σας. Η δυσκολία με τα δεδομένα είναι ότι μιλάμε για κάτι το πολύ πρόσφατο και εξορισμού δεν έχουμε τα δεδομένα γιατί δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να φορολογήσουμε. Δηλαδή είναι το γνωστό πρόβλημα, η κότα και το αυγό η ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Φορολογικού Συμβουλίου νομίζω είναι καλή και θα μας βοηθούσε ε, γιατί όπως είπε και ο κ. Κλίντ έχει τις πληροφορίες του, τις αναλύσεις του, έχετε τις δικές σας εσείς, έχουμε τις δικές μας εμείς, οπότε αξίζει νομίζω να έχουμε αντικειμενικά δεδομένα για να βασίζονται κάπου οι προτάσεις μας. Για τη μαύρη λίστα τώρα. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο επικριτικό. γιατί το γεγονό ότι έχουμε πέντε χώρε μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπου ε, Το ένα είναι ότι έχουμε πέντε χώρε, αλλά είναι, άρα είναι μικρό καταλόγος. Ε, το άλλο είναι έχουμε πέντε, ξεκινώντας από 17, άρα είμαστε αποτελεσματικοί. Εγώ αυτό θα έλεγα. Γιατί? Γιατί αποφασίζει βεβαίω ε, η ομάδα κώδικα συμπεριφορά, οπότε δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω. Αλλά αν δείτε το δικό μου το πρόγραμμα, το οποίο είναι δημοσίο. Και δείτε ποιοι, τους υπουργού οικονομικών από την γκρι λίστα έρχονται, ε, με επισκέφτονται, για να διορθώσουν την ομοθεσία τους, για να μην μπουν στη μαύρη λίστα. Και θα εκπλαγείτε πραγματικά. Μιλάμε λοιπόν για εντυπωσιακέ μεταρρυθμίσεις. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο στόχος της ε, μαύρης λίστας και γνωρίζω ότι υπάρχει νομίζω ακριβώς ε, το, υπάρχουν ελάχιστοι στη μαύρη λίστα του όσα και ακριβώς κάνουν προσπάθειες χώρες για να μην μπουν στην μαύρη λίστα και το θέμα είναι η γκρίζα λίστα όχι η μαύρη λίστα και δεν είναι κάτι το οποίο έγινε και τελείωσε είναι μια διαδικασία αυτό είναι το σημαντικότερο οπότε είναι σημαντικό να δούμε τι θα αποφασίσει η Επιτροπή αυτή του κώδικα συμπεριφοράς αρχές του 19 όταν θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις ε, δεσμεύσεις ε, οι οποίες ζητήθηκαν από κάποιες χώρες. Εάν ε, κάποιες δεν ακολουθούν τη σωστή προσέγγιση πρέπει να μπουν στη μαύρη λίστα. Εάν κάποιες αντιθέτως έκαναν κάτι πρέπει να βγουν από την μαύρη λίστα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι εν εξελίξη. Δεν έγινε άπαξ και τελείωσε και πιστεύω σε αυτήν την διαδικασία. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, συζήτηση αυτή και ήδη το είπαν κάποιοι συνάδελφοι ότι υπήρξε πρόοδος ε, στον τομέα κοινού ενδιαφέροντος ε, Κοινοβουλίου και Κομισιόν και ειδικά αν υπάρχει συμφωνία για την ψηφιακή φορολογία και για κάποια άλλα ζητήματα νομίζω ότι πραγματικά θα αφήσετε ένα μεγάλο κενό δυσαναπλήρωτο και το εκτιμούμε αυτό και δεύτερον συνειδητοποιώ ότι σας είχα ρωτήσει στις ακροά σα την ΕΚΟΝ για την σχέση σας με το Κοινοβούλιο και επιβεβαιώσατε αυτά τα οποία μας υποσχεθήκατε τότε και αυτό οφείλω να το πω και να είναι και ένα μήνυμα προς τους άλλους επιτρόπους ότι ο δρόμος επιτυχίας περνάει από το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ε, ίσως βοήθησε ότι ήμουν και δύο φορές Ευρωβουλευτής. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε σε λιγο

Well, let us, let Λοιπόν, ας ε, συνεχίσουμε με την δημόσια ακρόαση της Επιτροπής μας. Το κομμάτι αυτό αφορά τα συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και θα θυμάστε ότι η πρώτη τέτοια ακρόαση ήταν στις 21 Ιουνίου φέτος ε, με την συμμετοχή εκπροσώπων της McDonald's και της Nike. Σήμερα έχουμε την παρουσία εκπροσώπων του Group Caring, του Google, της Google και του Facebook. Οπότε καλώς ορίζω την κυρία Σοφή Μανταλώνη, υπεύθυνη φορολογίας στο group, στον Όμιλο Caring, τον κύριο Ανταμακόνο, επικεφαλής οικονομικής πολιτικής ε, στην αρμόδια περιφέρεια της Google και τον κύριο Άνταμ Λί, επικεφαλής παγκόσμιας φορολογικής πολιτικής στο Facebook. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως ε, με τις εισαγωγές, ε, τις τοποθετήσεις 7 λεπτών το πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν με την κυρία την κυρία Μανταλόνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές και μέλη της Επιτροπής. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που καλέσατε τον Όμιλο Κέρινγκ να μιλήσει στην Επιτροπή σας. Είμαι η Σοφία Μανταλόνη, είμαι διευθύντρια για τα θέματα, επιθυμητικά θέματα στον Όμιλο. Θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου κάνοντας μια παρουσίαση του ομίλου Κέρινγκ. Η Κέρινγκ είναι ο όμιλος ε, πολυτελείας ε, σε παγκόσμια κλίμακα. Μεγάλωσε ε, έχουμε διάφορους οίκους πολύ σημαντικούς του τομέα της ολογοπίας και της κοσμηματοπίας. Gucci έχουμε, Saint Laurent, Bottega Veneta, Valenciaga, Alexander McQueen, Μπριόνι, Bouchon, Πομελάτο, Dodo, Χιλίν, Ηλίς Ναρντά και Ζεράρ Περεγκού. Το 2017 ο Όμιλος Κέρινγκ είχε κύκλο εργασιών 15,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τη δημιουργία της το 1963, από τότε ο Όμιλας ε, συνεχώς μεταμορφώνεται, απασχολεί πάνω από 30.000 μισθωτούς, από αυτούς περίπου 16.000 στην Ευρώπη, και είναι παρόν όμιλο σε 46 χώρε μέσω ενό δικτύου 1.500 καταστημάτων, μπουτίκ. Για να σα παρουσιάσω λοιπόν τον όμιλο Κέρινγκ είναι σημαντικό ε, να αναφερθώ στη χρονολογία των διαφόρων βημάτων που οδήγησαν να γίνει όμιλο, όμιλος, όμιλος πολυτελείας, ε, κοινής ε, και πάντα ακολουθούμε επιχειρησιακή λογική στην νομική μας υπόσταση. Ο Φρανσουά Πινό μας ίδρυσε χρησιμοποιώντας υλικά κατασκευής και ξυλία. Είμαστε στον τομέα της διανομής από την δεκαετία των 90. Είχαμε το Printemps, La Redoute, την Conforama και τη Fnac στον Όμιλο. Η συμμετοχή, η ελεγκτική συμμετοχή στην Gucci Group που είχε συχθεί στη ΣΥΠΑ και στην Ολλανδία το 1993 σε 42% ποσοστό και αυτό ήταν ένα άλλο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του ομίλου και δημιουργήσαμε ένα σύνολο συνεκτικό και συμπληρωματικό των μεγάλων οίκων πολυτελείας. Αρχές του 2000 σημειώθηκαν από την απόκτηση οίκων του Yves Saint Laurent, του Sergio Rossi, της Bouchon, Bottega Veneta και Balenciaga που αγορίστηκε από την Gucci Group από το 2005 ε, επικεντρωθήκαμε εκ νέου στα προϊόντα πολυτελείας, ε, διανέμοντας στη Γαλλία τα προϊόντα και στην Ευρώπη, στο ευρύ κοινό. Μόνο από το 2011 και μετά η Gucci Group και η PPR συγχωνεύτηκαν και το 2012 η PPR έγινε μέτοχος 100% της του ομίλου Gucci. Το 2013 ο όμιλος PPR άλλαξε όνομα και έγινε Κέρινγκ. Πρώτο εξωτερικό σημάδι της μεταμορφώσεως. Έτσι, μέχρι το 2017 ε, έχει μόνο δύο αστηριότητες με τις οποίες ασχολείται. Τομέας πολυτέλειας και ε, τρόπου ζωής, lifestyle και ε, αθλητισμός και μέσα σε αυτό εντάσσεται το Πούμα. Το 2018 ε, ε, ξεκινά διαπραγματεύσεις με τη Στέλλα Μακάρτνεϊ Κρίστοφερ Κέιν και Τόμας Μάιερ για να τεθεί τέρμα στη συνεργασία μας. Ολοκληρώθηκε η μεταμόρφωσή μας και ασχοληθήκαμε μόνο με την πολυτέλεια έχοντας βγει από την Πούμα. Αλλά είναι μόνο το 2008 τα είδη πολυτελείας αποτελούσαν μόνο το 6% του κύκλου εργασιών. Στατηγική αλλαγή έγινε επιτυχής μόνο μέσω της επιχειρησιακής ε, προσέγγισης που ήταν αποτελεσματική. Η Κέρινγκ ανέλησε πολλά ζητήματα για να προσαρμοστεί επιχειρησιακά, για να παραμείνει ο οργανισμός σύγχρονος, ευέλικτος και να μπορεί να προσαρμόζεται σε έναν εκρηκτικό τομέα και εκρηκτική αγορά ε, έπρεπε να ασθενιστούμε νέου τρόπου κατανάλωσης, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ε, ηλεκτρονικό εμπόριο και ε, το, το μήλου Σανέλ μέσω των δικτύων αυτών. Χρειάστηκε εξυγχρονισμό. Ξεκινήσαμε το πρώτο εξάμεινο 2017 τον προβληματισμό, να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε όσον αφορά την ε, επιμελητία, τη διανομή ε, βασιστήκαμε σε ένα μοντέλο που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια. Περίπλοκο θέμα. Χρειάστηκε η παρέμβαση συμβούλων για στατηγική, για οργάνωση, για συστήματα πληροφορικής. Έτσι καταλήξαμε σε ένα σχέδιο ε, αλλαγής που επισημοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017. Μετά αυτή την αρχική φάση, μια νέα οργάνωση, διοργάνωση αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε χάρη στην οριμότητα των διαφόρων χαρτοφυλακίων του οίκου που προωθήθηκαν και, θέλαμε, και όλοι εργάστηκαν στον τομέα τους. Ε, λοιπόν, νέα οργάνωση, αναπτύξαμε προϊόντα, συντονιστήκαμε ε, και η παραγωγή, όλη αυτή η πτυχή ήταν ε, στα πλαίσια της κάθε μάρκας και στα κέντρα τεχνογνωσίας κάθε μάρκας. Βασιστήκαμε στις ανάγκες της επιχειρησιακές, και όχι σε φορολογικές πτυχές. Δεν επικεντρωθήκαμε σε αυτό. Η Κέρινγκ κινείται σεβόμενη τους εθνικούς φορολογικούς κανόνες και τις διεθνείς προδιαγραφές για τα φορολογικά. Και λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του ΩΣΑ ε, και λαμβάνει υπόψη και τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε νέα φορολογική οργάνωση εντός της οικονομικής διεύθυνσης. Τι μονατέθηκε. Και σε επίπεδο corporate και μάρκας είναι τα εξή. Πρώτα απ' όλα να ενοποιηθούν οι φορολογικές πληροφορίες σε επίπεδο μήλου ε, να παρακολουθούμε τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο σε τα φορολογικά, ε, να συμμορφωνόμαστε απόλυτα με την νομοθεσία, να εξασφαλίζουμε το σεβασμό των υποχρεώσεων που όσον αφορά την τεκμηρίωσή μας για τις συναλλαγές εντός μήλου, ε, να υπάρξει τεχνική συνεισφορά όσον αφορά τις πληροφορίες περιφορολογικών που αυτά θα λαμβάνονται υπόψη στους ενοποιημένους λογαριασμούς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχει καθορίσει η Γενική Διεύθυνση του Ομίλου για το θέμα αυτό. Ο όμιλο Κέρινγκ εκλήθη σε αυτή την ακρόαση, πως εκλήθη για να σας δώσει στοιχεία όσον αφορά τη φορολογική διακυβέρνηση που αποκλείει κάθε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Εν ονόματι του Ομίλου Κέρινγκ να σας παρουσιάσω ε, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε υπόψη τις εργασίες BEPS ε, στον φορολογικό προβληματισμό που ακολουθεί η ε, Όμιλος. Έχουμε στα πλαίσια του BEPS στόχο να εφαρμόσουμε τις αρχές της φορολογικής, της άμεσης φορολόγησης που υπάρχουν σε κάθε δικαιοδοσία. Ε, BEPS, κανόνε BEPS, αλλά να βάλουμε υπόψη και τη φορολογική μεταρρύθμιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, θέλουμε να μειωθεί η φορολογική, ο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ χωρών. Όσον αφορά τον όμιλο Κέρινγκ, μέσω παραδειγμάτων ε, κινούμεθα και θέλουμε να σας δείξουμε πώς εφαρμόσαμε τις στάσεις συλλογικά των BEPS χωρίς να αναλύουμε κάθε δράση BEPS. Ήδη έχουν ενσωματωθεί στο νομοθετικό σώμα ε, και στο ήπιο δίκαιο soft law. Η οικονομική μας διαχείριση ανταποκρίνει τις διεθνείς προδιαγραφές ε, όσον αφορά την διαμόρφωση των τιμών και είμαστε σίγουροι ότι οι εισφορές που καταβάλλονται εντός του ομίλου ευθυγραμμίζονται με σχετικούς κανόνες που αφορούν την τιμολόγηση και τις δραστηριότητες. Κάνουμε αναλύσεις λειτουργίας και κινδύνου συστηματικά και βαθμολόγηση ε, για όλους τους φορείς του ομίλου. Απόδειξη. Τι προσπάθειες κάνει η φορολογική διεύθυνση για αυτά τα θέματα και πόσο θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια όσον αφορά την τεκμηρίωση. Ε, ήδη αποφασίστηκε λοιπόν πάνω σε αυτό, πέρα από το local file και το master file, να παράγουμε και τεκμηρίωση για τις τιμές που διαμορφώνονται αναφορέα του ομίλου. Όσον αφορά την καταπολέμηση της καταχρηστικής χρήσεως των διαφόρων αποφάσεων και των συμβάσεων των φορολογικών, αποφασίσαμε ότι κάθε φορά που ένας φορέας της ομα... του ομίλου θέλει ε, να ε, ε, κινηθεί πρέπει να συμμορφώνεται κάθε φορέας με τις διάφορες αποφάσεις που υπάρχουν όσον αφορά την έδρα του κάθε οικού. Όσον αφορά την έννοια της σταθερής εγκατάστασης, της σταθερής έδρας, εφαρμόζουμε αυτόν τον ορισμό στον προβληματισμό μας για την εσωτερήκευση των δραστηριοτήτων μας του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το θέμα της σταθερής, του καθορισμού της σταθερής παρουσίας και της υπάρξης αποθέματος σε μια χώρα και της απόδειξης αυτού και τον επικουρικό και προποσχευαστικό χαρακτήρο, ε, τη ενία του νέου ορισμού, όλες αυτές οι πτυχές λαμβάνονται υπόψη. Τέλος, η ομάδα Κέρι δεν πει κανένα μέσο και δεν διαθέτει καμία υβριδική μονάδα. Ελπίζω ότι η εισαγωγή μου, ε, συγγνώμη που περεύει το χρόνο μου, θα συμβάλλει στην περαιτέρω συζήτηση και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στους ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόχαν από το Facebook. Σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εργάζομαι για... Είμαι επικεφαλής της οικονομικής ε, πολιτικής του Google για την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ασχολούμε τα τελευταία χρόνια με τα φορολογικά θέματα και έχω συμμετάσχει σε συζητήσεις με εθνικές κυβερνήσεις, τον ΟΣΑ, την Ένωση, διάφορες ομάδες ε, βιομηχανιών και επιχειρήσεων. Ήμουν εδώ το Μάρτιο του 2016. Η εταιρική φορολόγηση είναι θέμα έντονη συζήτηση ε, στην Ένωση, τις ΗΠΑ και αλλού. Και ο Σά και η Ένωση έχουν κάνει ε, αναλυτικές μελέτες. Και πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης θέλουν να εφαρμόσουν μια σειρά από αλλαγές στην πολιτική. Η Google από την πλευρά της πάντα ήταν υπέρ μιας πιο απλής και ε, συνεπούς φορολογικής πολιτικής. Όπως σας είπαμε από δύο χρόνια, η διεθνή μεταρρύθμιση στο φορολογικό τομέα θα επιτύχει μόνο αν οι επιχειρήσει έχουν σαφείς κανόνε και υπάρχει συνέπεια σε όλε τι δικαιοδοσίε. Είμαστε υπέρ τη πολυμερού προσέγγιση για οποιουσδήποτε νέου φορολογικού κανόνε, όπω αυτού που επιχειρούν να προωθήσουν το G20 και όσα εάν έχουμε μια κουρελού διαφορετικών κανόνων ε, από δικαιοδοσία σε δικαιοδοσία που θα αυξάνει τον κίνδυνο της διπλής ε, φορολόγησης και ε, παρατεταμένες δικαστικές διαδικασίες για φορολογικά θέματα θα έχουμε προβλήματα. Θέλουμε λοιπόν απλούς κανόνες και να μην υφίστανται διακρίσεις οι μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν εδώ και έναν αιώνα διεθνείς ε, συμβάσεις που προσπαθούν να δυσφαλίσουν την ε, ισότιμη μεταχείριση των ξένων εταιριών. Αυτοί οι κανόνες πάντα βοηθούν τα τελευταία δέκα χρόνια. Η Google έχει πληρώσει στην πράξη 26% φόρο. Πολύ παραπάνω από το 23,6% που είναι η υποχρεωτική φορολόγηση στις χώρες του ΩΣΑ. 6% από αυτό το φόρο πληρώθηκε στι ΗΠΑ, όπου ξεκίνησαν οι επιχειρήσει μα και όπου αναπτύσσονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίε μα. Τα υπόλοιπα πήγαν σε περίπου 50 χώρε στον κόσμο, όπου έχουμε μια σειρά από θηγατρικέ. Αυτή η κατανομή των φόρων μα ε, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι στοιχείο τη παγκοσμιοποιημένη οικονομία και ε, κανόνων για το πώς ε, πρέπει να φορολογούνται οι πολυεθνικέ επιχειρήσει αμερικανικές επιχειρήσεις πληρώνουν τον περισσότερο εταιρικό φόρο στη χώρα τους, όπως και οι γερμανικές, γαλλικές κτλ. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε έδρα στην Ιρλανδία, όπου έχουμε 8.000 ε, υπαλλήλου που παρέχουν υπηρεσίες παντού στην Αφρική, την Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Για να κάνουμε μια σύγκριση κλίμακα, έχουμε γύρω στου 40.000 μηχανικού στι ΗΠΑ που σχεδιάζουν και ε, παράγουν τα προϊόντα ε, που πουλάμε. Και έχουμε 3.000 μηχανικούς στην ε, Ευρώπη. Τώρα βέβαια άλλοι λένε ότι ο εταιρικό χώρος πρέπει να κατανεμηθεί διαφορετικά και να πάει από ε, τις χώρες όπου ε, παράγεται αξία α, περισσότερο στις χώρες όπου καταναλώνονται τα πρώτα και υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να το αποφασίσουν οι κυβερνήσεις, αλλά πρέπει να υπάρξει ευρία διεθνή συνένεση γι' αυτό, ούτω ώστε και οι κυβερνήσεις και οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Λί για το Facebook. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκπροσωπήσω το Facebook. Άλλαν Λί λέγομαι και είμαι επικεφαλής παγκόσμιας φορολογικής πολιτικής στην ε, Ουάσιγκτον. Ε, ήρθα στις ε, Βρυξέλλες από σεβασμό στο έργο της Επιτροπής σας και για να σας δώσω τις απαραίτητες πληροφορίες. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ στο επιχειρηματικό μας μοντέλο, τις επενδύσεις μας και τη συνεισφορά μας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Νομίζω ότι θα βοηθήσει να ξεκινήσω λίγο με το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Εμείς εξαρτώμεθα πρώτα απ' όλα από το να δημιουργούμε μια χρήσιμη εμπειρία στον χρήστη. 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 370 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, συνδέονται με το Facebook και τις άλλες εφαρμογές μας. 90% ε, των εσόδων μας προέρχεται από διαφημίσεις. Συχνά λοιπόν ε, ε, Βεβαίω, λογικό να εστιάζετε εσεί στη φορολογία. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στι επενδύσει τι οποίε κάνουμε. Θεωρούμε ότι το Facebook είναι ένα οικοσύστημα από τα προϊόντα τα οποία δημιουργούν οι μηχανικοί μα χρησιμοποιούνται για να ενισχυθεί η συνολική εμπειρία των χρηστών με το να ανεβάζουν αναρτήσεις, να συνδέονται με φίλους τους, να μπαίνουν σε ομάδες και να είναι σε επαφή με επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η διαφήμιση είναι ένα κομμάτι της εμπειρίας αυτής. Το να παρέχουμε μια τέτοια υπηρεσία για 2,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους είναι κάτι το σημαντικό συγχείρημα. Πέρσι το Facebook, όπως προκύπτει από τα στοιχεία μας, έκανε επενδύσεις κεφαλαίου 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σερβερ, κτίρια και υποδομές. Φέτος ήδη έχουμε ξεπεράσει αυτές τις υποδομές, έχουμε φτάσει στα 8,4 δισεκατομμύρια επιπλέον το Facebook δεν θα ήταν σε θέση να παρέχει την ε, εμπειρία αυτή χωρίς την καινοτομία. Και η επένδυσή μας σε έρευνα και ανάπτυξη έχει αυξηθεί ε, κάθε χρόνο. Ήταν 6,2 ε, δισεκατομμύρια ευρώ το 2017, αυξήθηκε από τα 5 δισεκατομμύρια το 2016 και βεβαίως παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές και σε επιχειρήσεις για να μπορούν να φτάσουν σε ένα νέο κοινό. Μάλιστα έχουμε κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις στην Ευρώπη πέρα από τα 17 γραφεία μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου απασχολούμε 7.000 άτομα έχουμε επενδύσει σε τέσσερα κέντρα δεδομένων, δύο ερευνητικά κέντρα σε τεχνητή νοημοσύνη και επιτρέψαμε σε πάνω από ένα εκατομμύριο μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αυξήσουν ε, τον τζίρο τους ε, και μιλάμε συνολικά για μια επένδυση 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη. Όσον αφορά τη φορολογική πολιτική, σε γενικέ γραμμέ είμαστε υπέρ απλών φορολογικών πολιτικών για τι επιχειρήσει που παρέχουν και σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Συμμετέχουμε σε διεθνεί τέτοιε συζητήσει και θεωρούμε ότι η συνεργασία μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων είναι η πιο αποτελεσματική, όπω θα θυμάστε ήμασταν ε, μία από τις εταιρείες που καταθέσαμε ενώπιον της Επιτροπής στο το 2015 και στον ΩΣΑ. Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει από την αρχική έκθεση του ΩΣΑ το 2014 η οποία κατέληξε ότι δεν θα είχε νόημα να διαχωριστεί η ψηφιακή οικονομία από την υπόλοιπη οικονομία για φορολογικούς σκοπούς. Εξάλλου, σιγά σιγά, η ψηφιακή οικονομία είναι κομμάτι της οικονομίας. Έκτοτε έχουν αλλάξει οι νόμοι και στις ΗΠΑ ε, οι οποίες ε, προχώρησαν προς ένα εδαφικό σύστημα όπως βλέπουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι ΙΠΑ υιοθέτησαν τις στάσεις του BEPS ε μαζί με κάποιους ελάχιστους συντελεστές πέρσι. Είπαμε ότι θα πάμε προς ένα μοντέλο τοπικών πολίσεων όπου το επιτρέπει ο νόμος και όπου έχουμε γραφεία και στον ΩΣΑ ακούμε συνεχώς πως θέλουμε να αυξηθεί ακριβώς η διαφάνεια για το πώς δημιουργούνται τα έσοδα αναχώρα. Αυτό κάναμε λοιπόν προληπτικά για να επιδείξουμε ακριβώ την προσήλωσή μα στον στόχο αυτόν. όπω βλέπετε είχαμε σημαντικέ αλλαγέ από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε πριν από τρία μόλι χρόνια. Η ικανότητά μα να επενδύουμε στην Ευρώπη βασίζεται σε ένα διεθνέ φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι απλό και θα παρέχει σταθερότητα σε όλε τι επιχειρήσει, ειδικά καθώ όλε οι επιχειρήσει πηγαίνουν προ την ψηφιοποίηση μα. ενθαρρύνει η συνεργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή εντό του ΩΣΑ και σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας μιλήσω και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οι ερωτήσεις θα γίνουν ως συνήθως σε μπλοκ των 5 λεπτών. Η κάθε ερώτηση ένα λεπτό το πολύ και ο υπόλοιπο χρόνος για απάντηση. Ξεκινάμε με τον συνεισηγητή από το ΕΛΚ τον κύριο Μάιερ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ δύσκολο να περιοριστώ στα 60 δευτερόλεπτα. Μιλήσατε, είπατε ότι θέλουν ε, απλούστερο, διαφανέστερο φορολογικό σύστημα επιχειρήσει. Πρέπει να είναι και βιώσιμο, θα τονίσω εγώ, και δίκαιο σε κάποιο βαθμό. Η πρώτη μου ερώτηση. Ξέρετε ότι ο ΣΑ εργάζεται στα πλαίσια ε, της ψηφιακής μόνιμης εγκατάστασης. Στην περίπτωση του Google και του Facebook, κατά την άποψή σα πώς είναι εφικτό να και οι δαπάνε και τα εισόδηματα να καταλογιστούν σε μια μόνιμη ηλεκτρονική εγκατάσταση στο μέλλον. Μετά, άλλη απληρώτηση. Ας πούμε ότι οι φίλοι μας πληρώνουν για μια διαφήμιση που κάνει Google ή Facebook και είναι, ο φίλος μου είναι στην ε, Τσεχία και έχει στόχο το τσεχικό κοινό, κατά την άποψή σας. Τα, τα κέρδη που θα παραχθούν από την ε, εταιρεία σας και ο φόρος που οφείλεται, πώς θα κατανεμηθεί στις διάφορες χώρες, πώς κατανέμεται τώρα, πώς θα έπρεπε να κατανεμηθεί και πώς κατανέμεται τώρα. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει, η Google. Με τα χαράς, ευχαριστώ για την ερώτηση. Θέλουν οι εταιρείε απλό, σαφές περιβάλλον φορολογικό, εύκολο να το διαχειριστούμε για την φορολόγηση των επιχειρήσεων Τώρα το πώς λειτουργεί το παρόν σύστημα. Η τεράστια πλειοψηφία των κερδών των εταιριών καταλογίζεται καταλογίζονται στην ε, τοπική αγορά. Το ίδιο και για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Θα οφείλονται τα περισσότερα κέρδη τους στη δική τους ε, αγορά. 66% παράγεται στη ΣΥΠΑ τα τελευταία 10 χρόνια και 14% στον υπόλοιπο κόσμο. Αν θέλουμε να γίνει ανακατανομή των κερδών και ποια φορολογικά δικαιώματα ανήκουν σε ποια δικαιοδοσία, πρέπει να συμφωνηθεί πολυμερό αυτό. Οι κυβερνήσει θα πρέπει να συζητήσουν και να αποφασίσουν πού θα εδρεύουν αυτά τα κέρδη. Η μεθοδολογία μέχρι τώρα ιστορικά βασιζόταν στη λειτουργία και κινδύνους που παράγεται στους διάφορους φορείς. Εμάς παράγονται βασικά στη ΣΥΠΑ. Μεγάλο ποσοστό αυτό αφορά την Ευρώπη και στην περίπτωση της Τσεχίας οι περισσότερες λειτουργίε εδρεύουν ε, στην Ιρλανδία. Και ο Τσέχος διαφημιστής ε, βασίζονται στην ε, υπηρεσία έρευνας αυτόματα σε βασικές ελέξεις κλειδιά σε επιχειρήσεις σε κάποια δημοπρασία χρησιμοποιούν τεχνολογία που παράγεται στην Καλιφόρνια και που ανεπτύχθη στην Καλιφόρνια ουσιαστικά. Όπως σας είπα έχουμε περίπου 40.000 μηχανικούς της ΕΠΑ και σχετικά μικρότερη παρουσία περίπου 3.000 στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, πρόσωπο τη Facebook. Παρόμοια απάντηση με του ίδιου κανόνες. Το κέρδος βασίζεται στους κινδύνους στοιχεία ενεργητικού δραστηριότητας και αυτοί οι κανόνες αλλάζουν και γι' αυτό γίνονται συζητήσεις στον ΟΣΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις νομές Είναι ευρύτερα ζητήματα περί κατανομής των κερδών. Αυτό είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων και θα πρέπει να υπάρξει συλλογική προσέγγιση, συνενετική με όλου του εμπλεκομένου. Θα πρέπει οι κυβερνήσει να συζητήσουν πού θα καταλογίζεται το κέρδο, πώ θα γίνεται η κατανομή των κερδών. Ευχαριστώ. Ο συνεισηγητής των σοσιαλιστών, ευχαριστώ πολύ που θα καταλογιζεται το κερδο πω θα γινεται η κατανομη των κερδων ευχαριστω ο των σοσιαλιστων ευχαριστω πολυ που ηρθατε στην ακρόαση. Ερώτηση για του εκπροσώπου Facebook και της Google. Αντιπροσωπεύετε από τις πιο, σε, τις πιο κερδοφόρες, πιο πλούσιες επιχειρήσεις στον κόσμο. Έστρεψε σε επαφή σχεδόν με κάθε πολίτη της Ευρώπης, τολμώ να πω καθημερινά, και βγάζετε κέρδος από αυτούς. Όχι μέσω τέλους, αλλά ουσιαστικά πουλώντας τους πρόσβαση Πουλώντα πρόσβαση σε αυτού μέσω προσωπικών πληροφοριών που διαθέτεται και μέσω πρόσβαση σε αυτού. Το Google έχει μεγαλύτερη αξία στην αγορά από ότι το ΑΕΠ τη χώρα μου, τη Δανία παράγεται αυτός ο πλούτος, όλο αυτό το κέρδος και πληρώνεται μόνο ένα κλάσμα των φόρων που καταβάλουν άλλες εταιρείες στην Ευρώπη. Η Facebook πέρσι είχα, σπάσατε ρεκόρ 1,5 δις ε, ευρώ στον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λιγότερο από 18 εκατομμύρια ευρώ πληρώσατε σε φόρους. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ πληρώσατε για δικαιτικές δαπάνες εντός εισαγωγικών. Πώς μπορούν οι διοικητικές σας δαπάνες να είναι πάνω από 27 πλάσιες από το ποσό που καταβάλλεται σε φόρους. Το Facebook το γι' αυτό και με το Google. Πέρσι πληρώσατε μόνο 55 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους για πωλήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι πωλήσει ήταν 6,5 δις ευρώ. Ερώτηση απλούστατα. Πώς γίνεται αυτό και πώς περιμένετε αυτά τα στοιχεία να αλλάξουν στο μέλλον, να εξελιχθούν στο μέλλον. Θα εξασφαλίσετε ότι θα καταβάλλετε τους φόρους απευθείας στις χώρες και τις κοινότητες ε, που βγάλετε τα κέρδη όχι μέσω ελλημοσύνης, αλλά πληρώνετε βάσει του ονομαστικού ε, φορολογικού συντελεστή της χώρας στην οποία έχετε παρουσία και που βγάλετε τα κέρδη. Πρόσωπος της Facebook 23% πληρώσαμε το 2017 4,6 δισεκατομμύρια σε φόρους. Υπάρχουν ευρύτερα ζητήματα που βρίσκονται ε, τα στοιχεία ενεργητικού που πρέπει να καταβηθούν οι φόροι. Συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες, συμμορφωνόμαστε με το ΩΣΑ, συζητούμε με τον ΩΣΑ και με εσά για να έχουν νόημα στο μέλλον οι κανόνες και να παράσχουν ε, κλίμα βεβαιότητας στις επιχειρήσεις. Για να διευκρινίσω κάτι που είπατε για την πώληση προσωπικών ε, στοιχείων. Δεν πουλάμε δεδομένα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και μετά χαρά συνεχίσουμε τη συζήτηση ποιοι είναι οι σωστοί κανόνες για κατανομή των κερδών. Ε, το εργατικό μας δυναμικό, συντριπτική πλειοψηφία είναι στην Καλιφόρνια, στο μέλλον πάρκ παράγεται το προϊόν και γίνεται και ο προγραμματισμός και η παραγωγή του προϊόντος στην Καλιφόρνια. Ε, το βάρος της Google ήταν 14,5 δολάρια Αμερικής η κατανομή του κέρδους και πού οφειλόταν ο μεγαλύτερο φόρο, κυρίω ο φόρος κατεβλήθη στη ΣΥΠΑ, 86% τα τελευταία 10 χρόνια. Ουσιαστικά έχουμε ένα σύστημα που κατανέμει τους, τα περισσότερα φορολογικά δικαιώματα εκεί που δημιουργούνται υπηρεσίες και τα προϊόντα και όχι εκεί που καταναλώνονται ε, δεν θα έπρεπε να αλλάξει ε, το σύστημα αν δεν υπάρξει συνεννόηση με τις κυβερνήσεις στον κόσμο. Αν κάποια κυβέρνηση πουν θέλουμε ένα σύστημα που βασίζεται στο που γίνεται η κατανάλωση και άλλο θέλει ένα σύστημα που βασίζεται εκεί που παράγονται και δημιουργούνται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα θα υπάρξει σύγκρουση στο διεθνές αυτό σύστημα. Ε, άλλη ερώτηση. Κοιτάξτε. Είπατε όπου γίνεται η κατανάλωση και παράγεται όμως και αξία από τους χρήστες για τις επιχειρήσεις σας. Είναι σαφές, δεν είναι μόνο κατανάλωση, αλλά παράγεται και αξία. Μετά, ρώτησα το Facebook και τα 500 εκατομμύρια ευρώ διοικητικών δαπανών στην Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι 17 φορές το ποσό του φόρου που πλήρωσε το Facebook στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι είδου δαπάνες είναι αυτές, μπορείτε αυτό ξεκαθέσετε, βέβαια απάντηση. Κόστος πωλήσεων, ουσιαστικά κόστος που αφορά τη λειτουργία των γραφείων μας, διοικητικές δαπάνες. Δεν δημιουργείται κέρδος και γι' αυτό πληρώνουμε φόρος. Ο φόρος εφαρμόζεται επί των κερδών. Ο διάλογος εκτός μικροφώνου. Αυτά είναι συνηθισμένα κέρδη που ε, ε, ε, σύμφωνα με τον νόμο. Κανονικά συζητούν οι χώρες για την κατανομή των κερδών. Και εμείς με τα χαρά σας μετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση, όπως προανέφερα. Πληρώσαμε 4,6 δις σε ευρώ σε όλο τον κόσμο. Αν υπάρξει αλλαγή, ε, αν θέλουμε να γίνει αλλαγή, με τα χαρά να το συζητήσουμε. Καλώς. Ευχαριστώ. εκπρόσωπος της Google για το θέμα της δημιουργίας αξίας. Ε, δεν πουλάμε δεδομένα των χρηστών. Οι υπηρεσίες μας δημιουργούνται και παράγονται στις ΕΠΑ και η προσθέμενη αξία ε, στις ΕΠΑ σημαίνει ότι και το κέρδος ε, εκεί πέρα προκύπτει. Και το ίδιο θα ίσχυε και για την ζημιά, αν υπήρχε ζημιά. Έχουμε θηγατρικές σε πολλές χώρες και στην Δανία που έχουν βεβαίως ε, με βάση τις ανάλογες ε, λειτουργίες και την σχετική κατανομή αλλά και τις ε, χρονιές όπου δεν είμαστε επικερδείς τοπικές εταιρείες πληρώνονται κανονικά, ενώ η μητρική εταιρεία στις ΗΠΑ υφίσταται και τις ζημιές και τα κέρδη. Οπότε αμφισβητείτε αυτό το οποίο είπα, λέει ο κ. Σκόφοντο, ότι δεν υπάρχει κάποια δημιουργία αξίας η οποία πρέπει να φορολογείται. Απάντηση. Τα δεδομένα των χρηστών είναι χρήσιμα για να κρίνουμε πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να δώσουμε το περιεχόμενο το διαφημιστικό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα οι αλγόριθμοι της αναζήτησης είναι το πολυτιμότερο κομμάτι του προϊόντος μας. Ε, αναπτύχθηκε στο Mountain View, χρησιμοποιεί μικρά κομμάτια δεδομένων για να δημιουργήσει έναν αλγόριθμο και τα περισσότερα δεδομένα που αφορούν ακριβώς την αναζήτηση είναι ένας κατάλογος ολόκληρου του διαδικτύου, όχι ε, τα δεδομένα των χρηστών. Ε, δηλαδή, τα δεδομένα του χρήστη είναι κατ' ουσίαν το ερώτημα που η αναζήτηση που μπορεί να ε, συγκριθεί με οποιαδήποτε καταναλωτική δραστηριότητα. ένα πολίτης ο οποίο μπαίνει σε ένα μαγαζί, ένας πελάτης, ο οποίο λέει θέλω να αγοράσω ένα ζευγάρι παπούτσια. Δηλαδή έχουμε ένα αίτημα για μια υπηρεσία και μια υπηρεσία η οποία παρέχεται. Η τεχνολογία όμως, η βασική και η τεχνογνωσία ε, αναπτύσσεται αλλού. Σας ευχαριστώ για το ΕΛΚ, ε, Ντάριος Ροζάτη. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μαντελενή και κύριοι καλώς ήρθατε. Να κάνω κι εγώ μία ερώτηση για το θέμα αυτό της δημιουργίας αξίας. Αυτό είναι το βασικό νομίζω και για τον καθορισμό του σωστού φορολογικού βάρους. Όπως αντιλαμβάνομαι η Google έχει 86% ε, των εσόδων ή των φόρων που πληρώνει στη ΣΥΠΑ. 86% του εταιρικού φόρου που πληρώσαμε τα τελευταία 10 χρόνια ήταν στη ΣΥΠΑ. Ανταποκρίνεται στο ποσοστό των εσόδων. Ο φόρος πληρώνεται στα κέρδη και όχι στα έσοδα και καμία πολυεθνική εταιρεία δεν θα έχει μια τέτοια αναλογία με άμεσο συσχετισμό του ποσοστού των εσόδων και του ποσοστού της ε, συνολικής φορολογίας. Ε, τώρα, επί σειρά ετών υπήρχε μια συζήτηση για αυτό το οποίο περιγράφεται, για μια κατανομή. Αλλά έτσι όπως λειτουργεί το διεθνές φορολογικό σύστημα αυτή τη στιγμή δεν βασίζεται σε αυτούς τους κανόνες. Δεν, δεν περιγράφω κάποιο σύστημα. Μία ερώτηση κάνω. 86% των κερδών των φόρων, μάλλον, 86% των φόρων καταβάλλονται στη ΣΥΠΑ. Φορολο... εταιρικής φορολογίας, όχι όλων των φόρων. Και 14% στις άλλες χώρες. Από κάποιες πηγές γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των χρηστών της Google είναι τουλάχιστον ο ίδιος με αυτό στη ΣΥΠΑ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αυτή η διαφορά στον φόρο που καταβάλλεται τι, είναι θέμα κόστους ε, το οποίο χρεώνεται στην πώληση ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη έτσι ώστε τα κέρδη σας ε, στην Ευρώπη να είναι τόσο λίγα ώστε και τα φορολογικά έσοδα μετά να είναι τόσο χαμηλά σε σχέση με τις ΣΥΠΑ. Νομίζω ότι αυτή η κατανομή του εταιρικού φόρου είναι φυσιολογική για οποιαδήποτε πολυεθνική όπως είπα και στην αρχή. Δηλαδή μια γαλλική ή γερμανική εταιρεία θα πληρώσει το, ε, τη μερίδα του λέοντος ε, της εταιρικής φορολογίας στην ε, μητρική της ας αγορά, στην, εκεί που έχει την εταιρεία της. Οπότε το σύστημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή φορολογικό παγκοσμίω βασίζεται στις λειτουργίες και στους κινδύνους των διαφόρων εταιριών. Όπως σας είπα στην Ευρώπη έχουμε 3.000 ε, μηχανικούς στην Ευρώπη και οπωσδήποτε υπάρχει εταιρική φορολογία. Είναι σαφώς λιγότερη από αυτή που καταβάλουμε στη ΣΥΠΑ. Κάποιοι συνάδελφοί μου έθεσαν το θέμα του ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε την ε, δημιουργία της αξίας ε, ως κάτι το οποίο δημιουργεί ο τελικός χρήστης. Εσείς έχετε διαφορετικό ορισμό από ό,τι φαίνεται. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πώς ε, δημιουργείται αξία εάν δεν έχετε χρήστες. Νομίζω καμία επιχείρηση δεν έχει έσοδα χωρίς πελάτες. Ναι, ναι. Αλλά όπως οποιαδήποτε επιχείρηση το θέμα Τη ε, εταιρική φορολογία είναι το πού δημιουργείται η αξία. Υπάρχουν άλλοι έμεση φόροι, διανομή κτλ. Ναι, ναι, αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Ε, δεν μιλάμε για την φορολογία των εσόδων όπως είπατε. Πράγματι όταν μίλησε για την ε, φορολογία των εταιρικών κερδών. Ναι, ναι, αυτό θέλουμε να ξέρουμε. Ποιο είναι ο μηχανισμό κατανομής που εξηγεί αυτή τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των κερδών που πληρώνονται στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη. Δεδομένου ότι ο αριθμός των χρηστών είναι λίγο πολύ ο ίδιο ή και υψηλότερο στην Ευρώπη. Ο μηχανισμός είναι μια γνωστή αρχή, λέγεται transfer pricing. Ε, υπάρχει σε διεθνείς φορολογικές συνθήκες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα του κόσμου εκτό διαδικτύου βασίζεται στις λειτουργίες και στους κινδύνους που αναλαμβάνει μια εταιρεία ή μια θηγατρική σε μια συγκεκριμένη αγορά. Γιατί χρησιμοποιούμε αυτή την αρχή. Γιατί θα έπρεπε να είναι ουδέτερο από φορολογική σκοπιά το πώς μια εταιρεία οργανώνει την λειτουργία της σε μια αγορά. Μπορεί να προσλάβει μια άλλη εταιρεία ή να δημιουργήσει μια δική της ε, δομή. Αυτό θα έπρεπε να είναι αδιάφορο από φορολογική σκοπιά και έτσι κατανέμονται τα κέρδη, δηλαδή καθορίζεται ένα ποσοστό κερδοφορίας ε, με βάση συγκρίσιμες εταιρείες που παρέχουν συγκρίσιμες υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ κύριε Κον. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Λί, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι, ε, τελειώνει ο χρόνος. Είναι παρόμοια ερώτηση. Είπατε ότι πληρώνετε 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ δολάρια στη ΣΥΠΑ με 300 εκατομμύρια τέλος δεν είναι όλοι που χρησιμοποιούν το facebook αλλά ας πούμε ίσως 250 εκατομμύρια χρήστες από την άλλη πληρώνεται 18 εκατομμύρια ευρώ φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο με πόσο ε, το 1 έκτο του πληθυσμού σύμφωνα με τους υπολογισμού μου Α, κατά κεφαλή πληρώνεται 15 ευρώ αναχρήστη φόρο στη ΣΥΠΑ ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 0,3 ευρώ αναχρήστη. Με άλλα λόγια, ε, σε μια παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή, το κόστος σας ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι πολύ υψηλότερο από ότι στις ΗΠΑ, γιατί στις ΗΠΑ έχετε πολύ μεγάλα κέρδη, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει κέρδο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχω τα στοιχεία για την υπόλοιπη Ευρώπη, απλά προσπαθώ να συγκρίνω τι δύο αυτές περιπτώσεις και θα ήθελα μια εξήγηση. Πράγματι ε, είναι ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Οι πελάτες μας είναι οι διαφημιστές, από εκεί έχουμε έσοδα. Και τα γραφεία μας ε, και οι εταιρείε μας ανά τον κόσμο κατά κανόνα υποστηρίζουν ακριβώς ε, τις πωλήσει αυτές. Πολλούμε διαφημίσεις σε διαφημιστές. Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αυτό το οποίο μου προξενεί εντύπωση είναι αυτή η τεράστια διαφορά κερδοφορίας ε, στη ΣΥΠΑ σε σχέση με τους χρήστες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, έχετε φοβερά, φοβερές διοικητικές δαπάνες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί δεν έχετε αυτό το κόστος στις ΗΠΑ. Κοιτάξτε, τα, να ξεκαθαρίσω, τα έσοδά μας είναι από τις διαφημίσεις και εκεί επιβάλλεται ο φόρος. Αυτή είναι η φορολογική βάση. Δεν ε, φτιάχνουμε ένα προϊόν το οποίο πουλάμε στους ε, καταναλωτές. Για τους χρήστες είναι δωρεάν ε, η υπηρεσία. Τα έσοδα είναι από τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές. Ωραία. Πολ Τάκ τώρα. Σοσιαλιστής. Σας παρακαλώ να είστε πιο σύντομοι γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους των εταιριών για την παρουσία τους. Τρεις ερωτήσεις. Αυτή η κατανομή ε, κερδών. Κυρίως ασχολούμαι με την Google και τη Facebook τώρα. Το εισόδημά σας κυρίως ε, καταχωρίζεται στην Ιρλανδία και για τις δύο εταιρείες σας. Ας ξεχάσουμε την κατανομή μεταξύ Ευρώπης και νομιμοντιών. Ας δούμε εντός της Ευρώπης έχετε λιγότερο από 5 εκατομμύρια χρήστες στην Ιρλανδία γιατί τόσο ο πληθυσμό. και έχετε περίπου 70 εκατομμύρια χρήστες στην Γερμανία αλλά το εισόδημά σας το καταχωρείτε στην Ιρλανδία και ε, πληρώνετε εκεί. Δεν καταχωρείτε εισόδημα στη Γαλλία τη Γερμανία. Είναι δίκαιο αυτό, το ότι δεν πληρώνετε τίποτα στη Γαλλία και τη Γερμανία. Γιατί οι χρήστε ε, είναι απαραίτητοι στο επιχειρηματικό σα μοντέλο. Δεν μπορείτε να λειτουργήσετε χωρί χρήστε. Δεύτερη. Ε, ε, έχω μια ιδέα για το τι θα απαντήσετε, αλλά τι, ποια είναι η γνώμη σας για τον ε, φόρο επί των ε, ψηφιακών υπηρεσιών. Και μια ερώτηση για τη Facebook. Αναφέρεται κάτι στην Επιτροπή Κελαφορών υπάρχει μία ε, προειδοποίηση για το εισόδημά σας σε σχέση με το φόρο. Σε σχέση με τις φορολογικές ε, αποφάσεις και κανονισμούς που έχετε σε διάφορες ε, χώρες. Ξέρω ότι έχετε θηγατρικές στη Δανία, τη Σουηδία και την Ιρλανδία είναι όμως και οι χώρες που είναι κατά του φόρου επί των ψηφιακών υπηρεσιών. Είναι σύμπτωση αυτό. Έχετε συμφωνίες φορολογικές στις χώρες αυτές. Και θεωρείτε ότι θα μπορέσουν να ισχύσουν επειδή έχουμε τις δραστηριότητες της κυρίας Φεστάγερ. Παρακαλώ. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγορών. Υπάρχει μια επιφύλαξη νομίζω. Μετά από κάποιο έλεγχο. Αυτές είναι συνηθισμένες ε, φορολογικές διαδικασίες ε, που μπορεί να ανεβάσουν, να κατεβάσουν το φόρο που πληρώνεις μια περίοδο. Οι φορολογικές ε, αποφάσεις και συμφωνίες είναι και αυτό το τμήμα της φορολογικής μας διαχείρισης. Δεν έχουμε ειδικέ τέτοιε αποφάσεις. Ε, διότι αυτές οι αποφάσεις δίνουν ασφάλεια και στους χρήστες. Επιτρέπει στις ε, φορολογικές αρχές να συζητήσουν με ένα φορολογούμενο οργανισμό. Δεν έχετε φορολογικές αποφάσεις. Στην Επιτροπή Φεραγωγών υπάρχει προειδοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια έρευνα σε διάφορες χώρες για το εάν και κατά πόσο δίδεται προτιμησιακή φορολογική συμπεριφορά μέσω κάποιων φορολογικών αποφάσεων, tax rulings. Έχουμε φορολογικέ αποφάσεις. Είναι φυσιολογικό τμήμα της ε, φορολογική μας διαχείρισης. Μπορεί να γίνουν έρευνε. Όχι, όχι, είναι μια τυπική ε, γνωστοποίηση. Τώρα για το θέμα του ψηφιακού φόρου. Θέλουμε να υπάρχει βεβαιότητα. Είναι θεμελιώδης αλλαγές του φορολογικού κώδικα. Οποιαδήποτε θεμελιώδης αλλαγή, για παράδειγμα η φορολόγηση του ακαθάριστου κύκλου εργασιών, για παράδειγμα, του, κύκλου, του ακαθάριστου εισοδήματο. Θα πρέπει να, να εισαχθεί με καλή προετοιμασία και συναντητικά. και η κατανομή του εισοδήματός σας ε, στην Ευρώπη. Είναι σωστό το ότι καταχωρείτε στην Ιρλανδία το εισόδημά σας που είναι τόσο μικρότερο από την Γαλλία και τη Γερμανία, όπου δεν καταχωρείτε εισόδημα. Το εισόδημά μας προκύπτει από τους διαφημιστέ. Και μετά τις συζητήσεις των ΟΣΑ και διάφορους ε, νομοθέτες όπως εσείς, έχουμε περάσει σε ένα ε, μοντέλο τοπικής παροχής υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι αυτό είναι πιο διαφανές. Αυτό ακούσαμε ότι λέτε εσείς που διαμορφώνετε την πολιτική και προς τα εκεί νομίζουμε ότι κινείται ε, η φορολογική πολιτική. Γκουα. Ο κύριος Μακάρθη. Ευχαριστώ. Τον εκπρόσωπο της Google τον ρωτώ τα για τη λεγόμενη διτή Ιρλανδική δομή. Στην τελευταία φορολογική δήλωση της εταιρείας Google Island Holdings που έχει έδρα το Δουβλίνου λέει ότι αυτή η διπλή που έχει η διπλή δομή Ιρλανδίας Βερμούδας που έχετε ε, εξακολουθεί να ε, ισχύει και από ό,τι ακούσαμε ε, η φορολογική σας έδρα είναι οι Βερμούδες Ακούσαμε διάφορα σχόλια. στο 2016 στη Βρετανική Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών ότι δεν έχετε ούτε έναν εργαζόμενο στη Φερμούδα. Ισχύει αυτό. Εξηγήστε μας τότε. Τι ωφέλη έχετε από τη συνεχιζόμενη χρήση αυτής της δομής. Μετά τη μεταρρύθμιση του φορολογικού κώδικα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης τα πνευματικά δικαιώματα στη Βερμούδα, τις Βερμούδες. Έχετε μετακινήσει πνευματικά δικαιώματα τα τελευταία δύο χρόνια από τις Βερμούδες στην Ιρλανδία και αν δεν το έχετε κάνει σκοπεύετε να το κάνετε. Επιπλέον, σε ποια δικαιοδοσία θα επάγονται τελικά τα πνευματικά σας δικαιώματα μετά το 2020. Ελπίζω ότι ήμουν συγκεκριμένος. Μια σειρά από ερωτήσεις. Να απαντήσω το πρώτο τελευταίο. Η δομή μας δεν άλλαξε. Τι συνέβη όμως στο παγκόσμιο προσκήνιο φορολόγηση, οι περικοπές, η νομοθεσία του, τον είπα άλλαξε για τη φορολόγηση και την απασχόληση πέρσι και επέβαλε ε, φορολόγηση όλες τις ιστορικά κέρδη ε, για αμερικανικές εταιρείες. Οι αμερικανικές εταιρείες αντίθετα πάλι πολυεθνικές ιστορικά έχουν φορολογηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι επί εδαφικού επίπεδου όπως οι άλλες μεγάλες ε, οικονομίες. Τι έκανε το σύστημα. Ανέβαλε τη φορολόγηση των διεθνών κερδών και όπως ε, ε, είπα και το 2016 στην Επιτροπή, η φορολογική δομή μα αντικατόπτρισε με αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματο των ΗΠΑ, που είναι μοναδικό. Και όλα αυτά λόγω του, νόμου που πέρσι θεσπίστηκε. Αυτά τα ιστορικά κέρδη φορολογήθηκαν. Αυξήθηκε η ευθύνη μα κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ για φορολόγηση στι ΗΠΑ το 2017. Ήταν ο φόρο και για το ρευστό και για τα στοιχεία ενεργητικού, ε, τα υπερπόντια. Και ουσιαστικά αμερικανική εταιρεία έχει την παροχή ε, των ε, υπηρεσιών, ο πάροχος των υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Έχουμε και την Google Island Holdings για την ανάπτυξη των πνευματικών δικαιωμάτων επί διεθνούς ε, επίπεδου. Σχεδιάστηκε αυτό για να αντικατοπτριστούν τα χαρακτηριστικά τα ιδιαίτερα του αμερικανικού φορολογικού συστήματος που άλλαξε θεμελιωδώς. Λοιπόν, σωστά το λέω όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ότι δεν έχετε καταχωρήσει κάποια πνευματικά δικαιώματα στις Βερμούδες. Όπως σας είπα, υπάρχει διεθέτηση συνειδιοκτησίας για τα πνευματικά δικαιώματα. Τελικά, η Alphabet Incorporated, που είναι η μητρική της Google LLC και των άλλων θυγατρικών, τα κατέχει. Θα μετακινηθεί, θα αλλάξει αυτή η διευθέτηση, θα μετακινηθεί από Βερμούδε σε άλλε δικαιοδοσίε συμπεριλαμβανομένω τη Ιρλανδία. Δύο παράγοντε παίζουν ρόλο. Είναι ε, η νομοθεσία περσινή για τη φορολόγηση των ΗΠΑ που άλλαξε και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται οι αμερικανικέ επιχειρήσει, ε, αυτέ που έχουν έδρα στι ΗΠΑ. Επίση, έχουμε τα συμπεράσματα BEPS του 2015, όπου εκεί βασικά τι είπαν, ότι οι εταιρείε τώρα θα πρέπει την ουσία και τη δομή των επιχειρήσεών του θα πρέπει να την ταιριάξουν με τη διεθνή δομή που είχαμε Εκεί εμπλεκόταν και οι Βερμούδε και η Ιρλανδία. Θα αλλάξει αυτό, σταδιακά θα εξαλειφθεί. Δεν ξέρω πώ θα γίνει αυτό. Την επόμενη διετία θα αλλάξει αυτή η δομή λόγω των αλλαγών BEPS που απορρέουν από το BEPS και όλων των αλλαγών που επέφερε, επέφερε το BEPS στην όλη δομή την ανάλογη της Ιρλανδίας τη φορολογική. Ευχαριστώ. Μαξ Άντερσον για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Ερώτηση. Έχω ερωτήσεις για τον όμιλο Κέρινγκ. Έχουμε πασίχνωστες μάρκες, Gucci, Φερρυπίν και Yves Saint Laurent. Και είχαμε και θηγατρική στην Ελβετία. Luxury Goods International LGI το όνομα αυτής. Αυτή η Luxury Goods International εισάγει ήδη πολυτελείας στην Ελβετία και ε, μετά τα αποθηκεύει και τα επαναπολεί τα προϊόντα σε υψηλότερο τίμημα, σε υψηλότερη τιμή σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει από δημοσιογράφους, η LGI πληρώνει μόνο 8% φόρο, πολύ λιγότερο από ότι είναι ο φόρος στις χώρες όπου τελικά βρίσκονται οι αγοραστές του προϊόντος. Αυτό είναι αρκετά κερδοφόρο. Η LGI παράγει μόνο 70% ε, της caring, παρόλο που απασχολεί μόνο 3% των υπαλλήλων που εργάζονται στον τομέα των ειδών πολυτελείας. Είπατε ότι ο όμιλός σας ε, δεν ε, ασκεί κανέναν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Τι αποκαλείται LGI, τι ονομάζεται LGI δεν κάνει φορολογικό σχεδιασμό. Τυχαίο είναι αυτό από πλευράς επιμελητίας και λογιστικών ε, υπολογισμών. 900 εκατομμύρια ήταν το καθαρό σας κέρδη, έκανε το LGI το 2016. Είδα τα στοιχεία στην ιστοσελίδα σας και το μέσο κέρδος εργαζόμενο στην Κέρινγκ είναι 13.000 ευρώ. Αρκετά καλό ποσό. Το μέσο κέρδος ανεργαζόμενο στην LGI είναι 1,5 δις. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Αν αυτό δεν είναι ένα κόλπο μετακίνησης ε, των κερδών και φοροαποφυγής, ούτως ώστε να μετακυλείτε, να μεταφέρετε τα κέρδη και να τα πηγαίνετε κάπου όπου οι φόροι είναι πολύ χαμηλά, τι είναι. Αν δεν είναι αυτό αποτελεί μετακίνηση ε, των φόρων, ε, των κερδών, συγγνώμη, που βρήκατε τόσο παραγωγικούς ε, εργαζομένους. Εσείς να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Η LG, η εταιρεία LGI, είναι κεντρικός κόμβος, hub, στα Caring. Δημιουργήθηκε εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Συναθρίζει διάφορες δραστηριότητες παρακολούθησης της παραγωγής, κάτι πολύ σημαντικό για τον Όμιλο, εποπτεία όσον αφορά την παραγωγή, έλεγχος παραγωγής, την επιμελητεία και τη διανομή. Εκεί επικεντρώνονται όλοι οι κίνδυνοι που διατρέχουμε όσον αφορά τη διανομή. Η LGI είναι ο χοντρικός πολιτής ομάδας, wholesaler. Είναι μια εταιρεία με 850 μισθωτούς. Πραγματική εταιρεία με επιχειρησιακή δραστηριότητα αδιαφυσβήτητη. Και μέχρι τώρα επέτρεψε την πρόθεση των μαρκών μας Χωρίς αυτό το κοινό εργαλείο, οι μάρκες μας δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθηκαν, χωρίς την LG. E. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι η LGI είναι ένα σύστημα που δημιουργήθηκε για φοροαποφυγή. Όλες οι μάρκες του μήλου είτε είναι κερδοφόρες είτε ελληματικές είναι εταιρείε που χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία, την πολύ μεγάλη τεχνογνωσία που έχουμε εντός αυτής της εταιρεία. τίποτα κύριε Άντερσον. Όχι. ΕΛΚ. Τόμ Φαντε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ακριβώς από πίσω σας. Θα απευθυνθώ και εγώ στην εκπρόσωπο της Κέρινγκ. Ε, Σε μια δήλωσή σας στο Reuters είπατε ότι μιλάμε για απτές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τώρα θα ήθελα να μάθω τι εννοείται ακριβώς με αυτό και απαντήσατε μόλις ε, στον κύριο Άντερσον. Γιατί όμως στην Ελβετία, τι κάνει την Ελβετία τόσο ελκυστική. Ε, υποθέτω ότι δεν είναι το μισθολογικό κόστος. Όσον αφορά το Facebook, ε, έχω μία ερώτηση για το local selling model, το τοπικό μοντέλο πολίσεων, το οποίο μοιάζει πολλά υποσχόμενο αλλά θα ήθελα να μου πείτε και εσείς ε, κάποια πράγματα ε, πώς ε, επιλέγετε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία το εφαρμόζετε. Παραδείγματος χάρη επηρέασε ακριβώ ε, την απόφασή σας να πάτε στο Ηνωμένο Βασίλειο το ότι χαμήλωσε ο φορολογικός ε, συντελεστής. Και τώρα από ό,τι κατάλαβα μιλήσατε για τοπική φορολογία. Για ποιου ποιους ακριβώς συντελεστές ε, μιλάμε και επίσης αν μπορείτε να μας πείτε και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτού του νέου μοντέλου φορολογίας. Σας ευχαριστώ κυρία Μαντελόνη. Παρακαλώ. Η ομάδα καταστάθηκε στην Ελβετία για λειτουργικούς λόγους. Η Σουηδία είναι στο κέντρο γεωγραφικά της Ευρώπης. Στρατηγική θέση γεωγραφικά για τα προϊόντα πολυτελείας. Τα προϊόντα μας παράγονται στη Γαλλία, την Ιταλία, που είναι κοντά λοιπόν στην Ελβετία, και η ευρωπαϊκή αγορά στην οποία απευθυνόμεθα όπως δημιουργήθηκε στις δεκαετίες 90 για λόγους λοιπόν γεωγραφικούς εγκατασταθήκαμε στην Ελβετία και για λόγους ασφάλειας έχουμε αποθηκευμένα προϊόντα που είναι ιδιαίτερα ακριβά και η Ελβετία μας έχει δώσει εγγύσεις ε, ασφάλειας για τα προϊόντα μας. Ο κύριος Λί. Κοιτάξτε, η δέσμευση και η δημόσια δήλωση που κάναμε ήταν ότι θα περάσουμε σε ένα μοντέλο τοπικών πωλήσεων όπου έχουμε ε, ένα γραφείο ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά από την Ευρώπη και μετά σιγά σιγά θα γίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μένουμε η διαδικασία αυτή που είναι πολύπλοκη και θέλουμε να γίνει σωστά και να συμμορφωνόμαστε με όλους τους τοπικούς νόμους αναμένουμε να κρατήσει δύο χρόνια τουλάχιστον. Όσον αφορά τώρα τους ε, φόρους και το ύψος, δεν μπορώ να το προβλέψω. Υπάρχουν ε, αλλαγές ε, που γίνονται τακτικά. Έχουμε δει πολλές τέτοιες αλλαγές, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι το μοντέλο αυτό θα καταλήξει σε μεγαλύτερο ποστό ρίσκου το οποίο θα πηγαίνει στην κάθε αγορά καθώς θα συμβάλλονται οι τοπικές εταιρείε με τους τοπικούς διαφημιστές. Θέλετε να κάνετε και άλλη ερώτηση. Ναι, σας ευχαριστώ. Έχω λίγο χρόνο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι είμαι ευγνώμων που ήρθατε εδώ. Ε, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να μας απευθύνετε μια επιστολή και το εκτιμώ που ήρθατε στην κυρία της ε, Κέρινγκ ε, τονίσατε την ε, σημασία της ασφάλειας για τα αποθέματά σας υπάρχουν. Νομίζω και ευρωπαϊκές χώρες όπου μπορείτε να φτιάξετε μια ασφαλή αποθήκη και για τον κύριο το Facebook σε ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε γραφεία. Uh, μπορώ. Δεν έχω πρόχειρο τον κατάλογο. Έχουμε 17 γραφεία στην Ευρώπη. Ε, μπορώ να τα... Έχουμε σίγουρα στο Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, στην Ιταλία, Ισπανία. Ε, μπορώ να σας στείλω τον, τον κατάλογο αν θέλετε είναι δημόσιες αυτές οι πληροφορίες. Ευχαριστώ να σας τις δώσω. Η ασφάλεια των αποθεμάτων προϊόντων μας είναι κάτι το θεμελιώδες. Ε, αυτά τα προϊόντα που έχουν αποθηκευμένα είναι το ενεργητικό μας, ε, ο πλούτος μας. Ε, υπενθυμίζω δεκαετία 90 όταν δημιουργήθηκε από το νόμιλο Gucci η υπήρχε μια χώρα πιο κοντά στην Ιταλία από ότι η Ελβετία που να μπορεί να παρέχει τέτοια ασφάλεια είναι εμφανές ότι η Ελβετία παρέχει ιδιαίτερη ασφάλεια είναι γνωστό ότι όλες οι εταιρείες ε, πολιτήμων λίθων και κοσμημάτων έχουν τα αποθέματά τους στην Ελβετία γιατί είναι πολύ ασφαλής. Πολύ ασφαλής για ε, αποθηκευμένα πολύτιμα προϊόντα. Εντάξει. Ολοκληρώνει το κατάλογο των ομιλητών μας. Πριν ολοκληρώσω, να ρωτήσω τους συνεισηγητές αν θέλουν το λόγο. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και τον τρόπο που προσπαθήσατε. Καταλαβαίνω ότι δεν σας ενθουσιάζουν οι ε, μονομερείς αλλαγές, αλλά ε, ε, κάτι πρέπει να γίνει από κοινού πρέπει να βρούμε ποιε είναι οι καλύτερε λύσει, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στο status quo. Δεν μπορούμε να το υπερασπιστούμε. Ελπίζω να συνεχιστεί η συζήτηση και να βρούμε μερικέ καλέ λύσει μαζί με διάφορε κυβερνήσει, γιατί μόνο μια συνολική λίστα είναι συνολική. Και εγώ σα ευχαριστώ και του τρει ομιλητέ για την παρουσία τους Ε, θα δούμε τις απαντήσεις, θα τις επεξεργαστούμε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το θέμα αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Έτσι ολοκληρώνεται η εργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Οι επόμενη συνεδριάσεις της Επιτροπής μας θα είναι στις 10 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο και στις 24 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Για τους συντονιστές και κλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση θα αρχίσει στις και μισή ακριβώς.